Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καθίστε παρακαλώ. Γιατί ήδη έχουμε δεκάλεπτη καθυστέρηση. Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο. Ας ξεκινήσουμε. Παρόλο που δεν είναι ακόμη όλα τα μέλη παρόντα. Ξεκινάμε όμως εμείς. Λάβατε το σχέδιο μέρησης διάταξης. της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης της 5ης 26 ε, Φεβρουαρίου για όλο ημέρη συνεδρίαση. Ερωτώ λοιπόν. Έχετε να προτείνετε κάποιες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Καταρχήν είχαμε μια έκτακτη συνεδρίαση των συντονιστών στο Στρασβούργο στις 11 Φεβρουαρίου και αποφάσισαν να ορίσουν οι συγητές για τέσσερα κατεπήγοντα θέματα. Είναι το σημείο 9-12 στην ημερήσια διάταξη. Η γραμματεία την περασμένη εβδομάδα μάλιστα σας έστειλε σχετικές ενημερωτικές πληροφορίες. Μπορούμε τώρα να εγκρίνουμε επίσημα τη συμπερίληψη και αυτών των θεμάτων στην ημερήσια μας διάταξη. Ευχαριστώ. Δεύτερον. <clears throat> Μετά τη δημοσίευση του σχεδίου στο σχέδιο σχέδιο διάταξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια καταξοδότηση πράξη. Μάλιστα ήμασταν υποψιασμένοι γι' αυτό ήδη από το Νοέμβριο του 2013 είχαμε το πρώτο σχέδιο αυτής της νομοθετικής πράξης και στις 19 Φεβρουαρίου την οριστική της μορφή. Αφορά τεχνικά μέτρα για προηγούμενες ε, πράξεις ώστε να ληφθεί ε, υπόψη η ίδρυση του νέου Ταμείου Αλίας και Θάλασσας και ο σχετικός κανονισμός. Στην Ολομέλεια του Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει ή θα απορρίψει αυτή την κατεξοδότηση πράξη μετά από σύντομη παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα αυτό θα είναι το τελευταίο σημείο της απογευματινής μας ημερήσιας διάταξης και στις 3 Μαρτίου 12 το μεσημέρι θα λήξει η προθεσμία για την ε, υποβολή της γνώμης μας για το θέμα αυτό. Συμφωνείτε να προσθεθεί και αυτό στην ημερήσια διάταξη. Θα είναι το τελευταίο σημείο της απογευματινής ημερήσιας διάταξης. Και τελευταία αλλαγή στην απογευματινή μας ατζέντα που θα είναι υπερπλήρης. Θα ήθελα να αλλάξουμε τη σειρά των θεμάτων 9 και 10 και των σημείων 11 και 12. γιατί Έχουν κάποια προβλήματα, έχει κάποια προβλήματα ο εισηγητή των σημείων 11 και 12. Λοιπόν, πρώτα θα συζητήσουμε το 11 και 12 και μετά τα 9 και 10. Συγγνώμη, εγώ είμαι εισηγήτρια μια έκθεση στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, η συνεδρίαση της οποίας συμπίπτει με τη δική μας απογευματινή. Και επειδή είμαι σκιώδη εισηγήτρια στο 9, Ε, δεν προλαβαίνω να είμαι παρούσα και στις δύο συνεδριάσεις. Δεν μπορούμε να το αναβάλουμε για άλλη φορά, γιατί είναι πολύ σημαντικό το 9. Είμαι σκιώδης ηγήτρια σε αυτό όπως σας είπα. Θέλω να μπορέσω να παρακολουθήσω τη συζήτηση και να λάβω το λόγο. Τέτοιες αλλαγές τελευταίες στιγμής ε, μας ε, δημιουργούν προβλήματα, γιατί συμπίπτουν δυστυχώς οι συνεδριάσεις πολλών επιτροπών και φροντίζουμε να οργανωθούμε εγκαίρως. Αν γίνονται αλλαγές τελευταία στιγμή, δεν προλαβαίνουμε να τα βολέψουμε. Ο κύριος Βανίλ Στερόι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με την αλλαγή των σημείων, αλλά επειδή υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, εσείς θα αποφασίσατε κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, δεν έχει έρθει ακόμα ο κύριος Μποστινάρου. Εκείνος ζήτησε την αντιστροφή των σημείων. Γιατί εκείνος είναι εισηγητής ε, στα σημεία 11 και 12 και με ειδοποίησε ότι πρέπει να φύγει νωρίτερα από τη συνεδρίαση γιατί έχει άλλες ενηλυμένες υποχρεώσεις και ζήτησε την αντιστροφή των σημείων. Ο κύριος Βανίστερ Ρόι είχε την καλοσύνη να δεχτεί αυτή την ε, αντιστροφή των σημείων. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν αντιρρήσεις. Αφού δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, θα παραμείνει αμετάβλητη η σειρά των σημείων παρά την ε, καλή διάθεση και την προθυμία του κύριου Βανίστερ Ρόι. Οπότε χωρίς την τελευταία αλλαγή εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και θα φροντίσουμε να τηρήσουμε το χρόνο μας και να προχωρήσουμε με καλή οργάνωση. Οπότε με τις αλλαγές αυτές που σας προανέφερα εγκρίνεται η μερίσια διάταξη και περνάμε στο σημείο 2, έγκριση των πρακτικών. Πρακτικά της συνεδρίασης ε, της 19ης και 20ης Ιανουαρίου. Ως συνήθως, αν μέχρι το τέλος συνεδρίασης δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένα τα πρακτικά. Εντάξει. Πολύ ωραία. Σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Μία σύντομη ανακοίνωση έχω μόνο. Έχετε λάβει ένα σύντομο ε, κείμενο σε κίτρινο, σε, συγγνώμη, σε άσπρο και κόκκινο. Ένα μικρό δωράκι από τη Βουλγαρία. Γιατί για τη Βουλγαρία η 1η Μαρτίου είναι πολύ σημαντική μέρα η 1η Μαρτίου. Είναι της γιαγιάς ε, Μάρθας ή της γιαγιάς του Μαρτίου. Και είναι η μέρα που ανταλλάσσουμε ευχές ε, υγείας, για καλή υγεία, για επιτυχία, για τύχη και βάζουμε και αυτή την ε, ασπροκόκκινη αλυσιδίτσα, το Μάρτι που λέμε και στα ελληνικά. Αυτό το δωράκι λοιπόν από την Πρόεδρο. Και περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, την επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη την πρόθεση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση. Αυτό είναι το πρώτο ουσιαστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, πρόκειται για την έκθεση που αφορά την έκτη έκθεση συνοχής ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε τρία χρόνια υποβάλλεται η έκθεση για την ε, συνοχή. Τον περασμένο Ιούλιο υπευλήθηκε η τελευταία έκθεση συνοχής για την πολιτική συνοχής 2007-2013. Μετά τις ε, σημαντικές περικοπές της δημόσιας επενδύσεις ε, λόγω κρίσης και αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων εξετάζεται η συνέπεια στην ε, πολιτική συνοχής. Η δημόσια υποστήριξη περνάει από θέματα μεγάλων υποδομών σε θέματα ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης ε, και στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Δεκέμβριο ο εισηγητής μας ο κύριος Ντόιτς μας παρουσίασε τις ε, πρώτες του σκέψεις για το περιεχόμενο της ε, έκθεσης και σήμερα θα μας παρουσιάσει το πρώτο του σχέδιο έκθεσης. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών λίγη την 5η 12 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στις 15 Μαΐου στην Επιτροπή στις 5 συγγνώμη Μαΐου στην Επιτροπή μας επί της εκθέσεως και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ντόιτς να σας αναφέρω ότι έχουμε και εκπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών στην συνεδρίασή μας τον Σένα Άλμπερτ Πόρτ που θα μας παρουσιάσει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών. Έχουμε εκπρόσωπους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Ο κύριος Παύλο Μπάρος Βάλλη είναι ο αρμόδιος συγητής της ΟΚΕ. Πρέπει να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι με το χρόνο. Ε, όπως σας είπα είναι υπερφορτωμένη η μερίσια μας διάταξη. Γι' αυτό και θα δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ντόιτς. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, συζητά σήμερα την έκτη έκθεση συνοχής ή τουλάχιστον το σχέδιο γνωμοδότησης το δικό μου επί του ζητήματος. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων επ' αυτού. Θα ήθελα καταρχάς να σας υπενθυμίσω τα τρία ουσιαστικά σημεία που αποτελούν και τη βάση της γνωμοδότησής μου. Η Πρόεδρος ε, ήδη αναφέρθηκε στα σημεία αυτά και τα έχουμε συζητήσει άλλωστε Καταρχάς, ε, νομίζω ότι είναι θεμελιώδη σημασίας ε, το γεγονός ότι τα προβλήματα ρευστότητας θα πρέπει να επιληθούν. Γι' αυτό και στο σχέδιο γνωμοδότησης επικεντρώθηκα στο θέμα αυτό. Η καθυστέρηση πληρωμών είναι περίπου 25 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Γεγονός το οποίο είναι εις βάρος της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής. Στο σχέδιο έκθεσης λοιπόν ε, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ένα θεματολόγιο το οποίο θα περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό φέτος το 2015 να μπορέσουμε ε, να έχουμε κάποια βήματα και ε, να ε, υπάρξει κάποια αρρύθμιση όσον αφορά τις καθυστερήσεις. Θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσει η διαδικασία για το 2014-2020 έχουν υποβληθεί 387 προγράμματα, από τα οποία εγκρίθηκαν τα 266 και είναι απαράδεικτο να βρισκόμαστε πλέον στην άνοιξη του 2015 και να, έχουμε μόνο το, να έχει περάσει το 20% δηλαδή του αρχικού διαστήματος και τα επιχειρησιακά προγράμματα να μην έχουν ακόμα ξεκινήσει. Το 1 τρίτο αυτών των προγραμμάτων δεν έχει καν εγκριθεί. Στο σχέδιο γνωμοδότησης λοιπόν ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, ε, ε, εξηγήσει λίγο τις αναμενόμενες οικονομικές συνέπειες αυτής της καθυστέρησης και θα ήθελα να προτείνω επίσης να μας πούνε και πώς σκοπεύουν να διορθώσουν αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Σε γενικές γραμμές η σχέση με την ε, στρατηγική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντική και την τονίζω εδώ στη γνωμοδότηση. Η πιο σημαντική πολιτική επενδύσεων, η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της παρούσας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε η πολιτική συνοχής να θεωρηθεί απλώς ένα εργαλείο, ένα μέσο για την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Το άρθρο 174 της Συνθήκης προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλίσει ε, την ε, απρόσκοπτη ανάπτυξη θα πρέπει να βελτιώσει την παραγωγικότητά της ώστε να διασφαλίσει κοινωνική, οικονομική συνοχή και να μπορέσει να μετριάσει τις δυσκολίες ε, ε, που προκύπτουν λόγω των διαφορών ε, στο επίπεδο ανάπτυξης των διαφορών περιφερειών. Γι' αυτό και ακριβώς εγώ στη γνωμοδότησή μου εφιστώ την προσοχή στο γεγονός ότι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τον αρχικό στόχο της πολιτικής συνοχής ε, ο οποίος είναι γεγραμμένος και στη συνθήκη, ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική συνεισφορά στην παρούσα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο βασικό στοιχείο της νομοδότησης είναι κάτι το οποίο έχω αναφέρει και στο παρελθόν, είναι το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Δεν αρκεί να μένουμε στην ε, αποτελεσματική εφαρμογή της ε, προγραμματικής περίοδου 2014-2020, θα πρέπει να δούμε και το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Ιδάλλως, το 2019 θα βρεθούμε αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα. Οι νέες πολιετές δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την πολιτική συνοχή και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προετοιμασία και ε, ε, του νέου κύκλου συγγνώμη, πολιτικής συνοχής. Γι' αυτό ακριβώ και θα πρέπει να ξεκινήσει ήδη η διαδικασία εξέτασης της μελλοντικής πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Πέραν αυτών των τριών ουσιαστικών στοιχείων υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία τα οποία επισημαίνει η έκθεση και θα ήθελα να σας ε, τα αναφέρω συνοπτικά. Να ξεκινήσω με τη σχέση μεταξύ του πακέτου Juncker και της πολιτικής συνοχής. Η γνωμοδότησή μας για το πρόγραμμα επενδύσεων θα συζητηθεί σήμερα το απόγευμα εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά θα ήθελα να αναφέρω εδώ στο σχέδιο γνωμοδότησης ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε και σχέση μεταξύ ε, των ε, διαθροτικών ταμείων του Ταμείου Ανάπτυξης και του πακέτου Juncker. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται μια κοινή πολιτική συνοχή, η οποία θα είναι ευθυγραμμισμένη με το σχέδιο το οποίο έχει προτείνει ο κ. Γιούνκερ. Η πολιτική συνοχής και ο σχετικός προϋπολογισμός δεν μπορούν να περιοριστούν λόγω του πακέτου Γιούντερ και στα πλαίσια της εφαρμογής του πακέτου θα πρέπει να ε, δούμε και τι γίνεται με την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης που ξεκίνησε το 2008 και να χρησιμοποιήσουμε και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα. Υπάρχει ένα επίπεδο μόχλευσης και πολλαπλασιασμού το οποίο φυσικά είναι πρόσδεκτο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να πλουστεύσει τη χρήση των ε, διαφόρων χρηματοπιστωτικών μέσων. Η κρίση μας έχει αποδείξει ότι η πολιτική συνοχής δεν είναι απλώς χρήσιμη, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να απαρνηθούμε είναι μια ευρύτερη πολιτική που έχει αποδείξει ε, και πόσο ισχυρή είναι. Ε, η κρίση όμως μας επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι ε, είναι, η συνοχή είναι ένα στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να προσταθούμε περισσότερο στην εφαρμογή του επόμενου κύκλου. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αναφέρω και τρία πράγματα. Καταρχάς ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να είναι αποτελεσματικές επενδύσεις στη συνοχή. Αλλά οι όροι της μακροοικονομικής αρεσιμότητας θα πρέπει να εφαρμόζονται εδώ. Και εδώ το Κοινοβούλιο ε, θα ήθελε να λαμβάνει αγκαίρους πληροφορίες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και φυσικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αποτελεσματική επιτροπή ε, εφαρμογή συγγνώμη σαφώς είναι ευπρόσδεκτη, αλλά χρειαζόμαστε και κατάλληλες πολιτικές για τις διάφορες περιφερειακές για να λάβουμε υπόψη και τις διάφορες τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών είναι κάτι που θα μπορούσε επίσης να συνεισφέρει για να μειωθεί το επίπεδο ασφαλμάτων και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και το θέμα της απασχόλησης είναι κάτι το οποίο ε, αναφέρεται ε, και τονίζεται στο σχέδιο γνωμοδότησή μου. Η κρίση έχει πλήξει την ε, αγορά εργασίας και επομένως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει κατάλληλη ένταξη και στην αγορά εργασίας αλλά και στην κοινωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά εάν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και να υπάρχει και κατάλληλη υποστήριξη από το ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εγώ λοιπόν ε, υποστηρίζω την ολοκληρωμένη χρήση αυτών των ταμείων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επομένως χρειαζόμαστε ε, νομοθεσία και διοικητικές διαδικασίες οι οποίες θα διευκολύνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για τη λήψη χρηματοδότησης και για τη μείωση του περιτού γραφειοκρατικού άχθους. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, ανάπτυξη επίσης ε, επιχειρησιακών δεξιοτήτων για να μπορούμε να ενισχύσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μας ανησυχεί επίσης ιδιαίτερα το γεγονός ότι η ενεργεία των νέων είναι άνω του 20% στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι είμαστε σε διπλάσιο ποσοστό ε, σε σχέση με τους, το σύνολο των ενηλίκων ανέργων. Επομένως θα πρέπει να κινητοποιήσουμε κονδύλια το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να υποστηρίξουμε ε, την απασχόληση των νέων ανθρώπων. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε επίσης σε ευάλωτες ομάδες, άτομα με αναπηρία, άτομα ε, με ε, κοινωνικές ή άλλες μορφής αναπηρίας. Και θα ήθελα να αναφερθώ και στην εδαφική διάσταση, η οποία δεν έχει λάβει την προσοχή που της αξίζει. Η εδαφική συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο προκειμένου να βελτιώσουμε την κινητικότητα στην αγορά εργασίας, την ανάπτυξη του τουρισμού και ούτε καθεξής. Πρόκειται για θέματα στα οποία είναι πολύ σημαντική και η διασυνοριακή διάσταση. Η εδαφική ανάπτυξη είναι κάτι περίπλοκο, το οποίο θα πρέπει να βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και τις σχετικές ομάδες ε, Υπάρχει ο Ευρωπαϊκό όμιλο Εδαφική συνεργασία και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη της υπαίθρου και την ε, πολιτική συνοχή εδώ. Η νομοθεσία για την ε, πολιτική συνοχή και ο σχετικό κανονισμός βασίστηκαν σε ευρεία κλίμακα συντονισμό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ε, καταλήξει σε μια κοινή θέση. Όσον αφορά την έκτη έκθεση για τη συνοχή, ε, πρόκειται για μια ευκαιρία για να ανανεώσουμε και να δώσουμε μια νέα όθηση στην πολιτική συνοχή. Γι' αυτό και ακριβώς στόχος μας είναι μια κοινή πολιτική θέση. Πρέπει να συζητήσουμε τον κοινωνικό και οικονομικό ρόλο της πολιτικής συνοχής, πρέπει να συζητήσουμε τις προκλήσεις, καθώς επίσης και ε, τι σκοπεύουμε να κάνουμε προκειμένου να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα. Πρέπει να δούμε και το μέλλον και τις προοπτικές μετά το 2020. Εγώ είμαι αισιόδοξο ε, για την συνεργασία μας. Υπήρξε πολύ καλός συντονισμός ε, με τους κοιόδη συντάκτες μέχρι τούδε και ε, φυσικά προσβλέπω και στις απόψεις σας για το σχέδιο γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Yes, uh, thank you. Ευχαριστούμε κυρία Μπρεσό από τους σιώδης συγητές, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Ντόιτς, ο οποίος μας παρουσίασε μία έκθεση πλήρη και με την οποία σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε κυρίως όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Συμφωνώ επίσης πλήρως, αλλά νομίζω ότι και όλη η Επιτροπή μας ε, θα συμφωνήσει, διότι έχει υπάρξει και σχετικό ψήφισμα για το θέμα της καθυστέρησης των πληρωμών, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό για τις περιφέρειες και τις πόλεις μας και κυρίως για τους χρήστες της πολιτικής συνοχής. Κατά την άποψή μου, είναι λίγο πιο αδύναμη ανάλυση όσον αφορά το παρελθόν δηλαδή την ανάλυση που σχετίζεται με τα ισχυρά στοιχεία και τα κενά σε σχέση με το παρελθόν, ο συνάδελφος επικεντρώθηκε πρωτίστως στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω 4-5 παρατηρήσεις ε, για την έκθεση, οι οποίες θα μπορούσαν ίσως να χρησιμεύσουν για την ανάλυση για το μέλλον. Πρώτον, ανακύπτει εκ νέου το θέμα της ε, βελτίωσης της ποιότητας της δημόσιας δαπάνης. Ε, με πολλές δυσκολίες καταφέρνουμε να δαπανίσουμε τους πόρους μας, αλλά δεν είναι πάντα ποιότητα ποιότητας δαπάνη. Και, και σε αυτή την έκθεση, παρά το γεγονός ότι πάντα λέγεται ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τα αποτελέσματα, ε, αποτελέσματα και με ποιοτικούς όρους, ε, πολύ συχνά αυτό που κάνουμε είναι να περιοριζόμαστε απλώς ε, στη ε, δυνατότητα να δαπανίσουμε κονδύλια. Θα πρέπει να προσέξουμε λίγο καλύτερα τα αποτελέσματα γιατί εδώ είναι λίγο αδύναμο το κείμενο. Ένα θέμα το οποίο προκύπτει σαφώς στην ανάλυση των πινάκων και των στοιχείων και των διαγραμμάτων που μας δίνεται είναι ότι υπήρχε μία τάση να επικεντρώνονται οι πόροι σε περιφέρειες και πρωτεύουσες και αυτό είναι προφανέστατο ακόμα και σε χώρες που είναι χαμηλότερου δήματος. Πάντα οι πρωτεύουσε ε, βρίσκονται στην κορυφή, ξεπερνούν ε, ακόμα και το 100% του ευρωπαϊκού μεσοόρου, ενώ οι περιοχές της Υπέθρου αλλά και οι, περιοχές, ε, και οι πόλεις των πιο περιφερειακών περιοχών που δεν είναι απαραίτητο μικρές αλλά είναι πιο περιφερειακές δεν έχουν αντίστοιχα τόσο μεγάλη ανάπτυξη. Ελοχεύει λοιπόν ο κίνδυνος να δημιουργηθούν ε, διαφορές ή να ενταθούν οι διαφορές εντός και των ίδιων των ε, κρατών. Κάτι επιπλέον σε σχέση με το παρελθόν οι διαδικασίες ε, κυρίως ε, για τη χρήση των κονδυλίων της πολιτικής ε, συνοχής και κυρίως για τα μέσα της, τα χρηματοπιστατικά είναι ιδιαίτερα επαχθείς και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Επειδή στην επόμενη προγραμματική περίοδο προβλέπεται μια πολύ μεγαλύτερη χρήση των χρηματοπιστωτικών μέσων, κάτι το οποίο με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη, θεωρώ ότι θα έπρεπε να διευκολύνουμε λίγο τη χρήση τους και να είναι πιο απλά. Ένα τελευταίο για το παρελθόν. Η οικονομική κρίση Ε, κατέδειξε ότι ένα διάστημα 7 ετών είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ένας προγραμματισμός που είχε γίνει πριν από την κρίση έπρεπε να ε, περάσει στην εφαρμογή του και στη διαχείρισή του εν μέσω κρίσης και αυτό δημιούργησε ένα μεγάλο αριθμό επιπλέον κανόνων. Ε, πλέον οι οικονομικοί χρόνοι επιταχύνονται ολοένα και περισσότερο. Επομένως θα πρέπει να προβλέψουμε μία ε, πιο στεναρή μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, η οποία θα μας επιτρέπει, ε, θα επιτρέπει μάλλον στα κράτη και στις περιφέρειες να προσαρμόζουν τον προγραμματισμό τους ανάλογα ε, με τις ολοένα ε, κειμενόμενες οικονομικές συνθήκες. Μια μεγαλύτερη λοιπόν ευελιξία στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, ώστε να αποφύγουμε ακριβώς να βρισκόμαστε ενώπιον του ίδιου κινδύνου, να μην είμαστε συντονισμένη με τις συγκυρίες. Όπως σας είπα, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις παρατηρήσεις του συναδέλφου, ιδίω όσον αφορά την μακροοικονομική ε, διάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αν αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Το Κοινοβούλιο ήταν πάντα κατά της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, ε, και το, αλλά αν αποφασιστεί να χρησιμοποιηθεί, τότε θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συμμετέχει προκειμένου να αξιολογήσει αν είναι σωστό να χρησιμοποιηθεί ή θα είναι κάτι που θα επιδενώσει ίσω την κατάσταση αντί να τη βελτιώσει στα κράτη-μέλη. Συμφωνώ απολύτω λοιπόν με την παρατήρησή σα αυτή. Δεύτερον, να συμφωνήσω επίσης ε, και ε, με την παρατήρηση και θα το συζητήσουμε και σήμερα το απόγευμα ε, για την ανάγκη συντονισμού μεταξύ του σχεδίου Juncker και της πολιτικής συνοχής. Σίγουρα δεν πρόκειται για το ίδιο πράγμα, αλλά επειδή έχουν γίνει και θα γίνουν μεγάλες προσπάθειες επενδύσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης επ' αυτών των δύο, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ε, θεματικές ενότητες και θα πρέπει να δώσουμε και τη δυνατότητα στα κράτη, στις περιφέρειες και στις πόλεις να έχουν ένα κοινό συντονισμό και να δημιουργηθεί συνέργεια μεταξύ των διαφόρων μέσων. Τρίτον, όπως σας είπα και προηγουμένως και ισχύει φυσικά και για το μέλλον, Πάμε όλο ένα και περισσότερο προς ε, ε, χρηματοπιστωτικές ε, τεχνικές και επομένως μια απλούστερη διαδικασία και μια πιο εύκολη εφαρμογή τους θα δημιουργήσει μέσα τα οποία θα είναι πιο ελκυστικά. Κάτι τελευταίο όσον αφορά τα νέα μέσα προγραμματισμού, τα οποία όπως γνωρίζετε εγκρίθηκαν με κάποια καθυστέρηση λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται κυρίως με την ιστέρηση ε, στην ε, έγκριση του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Εδώ η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει πολύ επικίνδυνη για τις περιφέρειες, διότι μπορεί να τους ζητηθεί να χρησιμοποιηθούν τους πόρους δύο, ή πόροι δύο ετών 2014-2015 μόνο εντός ε, του έτους 2015. Και ο κίνδυνος είναι ε, για πολλές περιφέρειες ο χρόνος αυτός να περιοριστεί σε λίγους μήνες γιατί η τελική έγκριση θα δοθεί την άνοιξη ε, αν όχι και αργότερα και τελικά μέσα σε ένα εξάμεινο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο χρόνια προγραμματισμού. Το να επιτρέψουμε ίσως να τα απλώσουμε λίγο καλύτερα. Σε δύο χρόνια προγραμματισμού τη χρονιά που χάθηκε διότι δεν ήταν και δική τους ευθύνη κατά την άποψή μου θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, διότι ελοχεύουν να υπάρχουν καθυστερήσεις στις δαπάνες και μάλιστα ε, ε, ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Στην ε, παρουσίαση του κυρίου Ντόιτς ε, δεν νομίζω ότι άκουσα κάποια αναφορά στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές είναι μια πραγματικότητα που συνδέεται όλο και περισσότερο με την πολιτική συνοχή και επομένως ε, φρονώ ότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην επόμενη έκθεση ε, θα πρέπει να γίνει μία ανάλυση του πώς οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές της μακροπεριφέρειες χρησιμοποιούνται ή δεν χρησιμοποιούνται, αν χρησιμοποιούνται με συντονισμένο τρόπο, αν συνάδουν με τα εγκεκριμένα προγράμματα, με τους ε, πόρους της πολιτικής συνοχής και αυτό θα ήταν χρήσιμο. Ε, από εκεί και πέρα θα δούμε κατά πόσον θα πρέπει να υποβληθούν τροπολογίες, αρκεί να υπάρχει μια μηνύα η οποία θα λέει ότι θα θέλαμε στην επόμενη έκθεση κάποιες ενδείξεις, κάποια στοιχεία για την ε, εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και κατά πόσον πραγματικά συντονίζονται με την πολιτική συνοχή. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μπρέσο. Η κυρία Τόμασιτς που είναι σκιώδης συγγετρία. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας τον κύριο Ντόιτς για την πολύ αξιόλογη του έκθεση. και τις πολύ χρήσιμες συστάσεις του για τη μελλοντική πολιτική συνοχής. Για την περίοδο 2014-2020 θα περάσει μεγάλη μεταρρυθμίση ρηξη και έλευθη για να ενισχυθούν οι σχέσεις της, ε, της ε, πολιτικής συνοχής με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συνδυαστεί η αποτελεσματικότητά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια ολοκληρωμένη σφαιρική προσέγγιση και αυτό να είναι ο κανόνα. Έτσι θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στην αποτελεσματικότητα και στην υλοποίηση των στόχων, αξιοποιώντα καλύτερα τι επενδύσει. Έχουμε πολύ περίπλοκες προκλήσεις για τις περιφέρειες και θα πρέπει να θετήσουμε ένα συντονισμένο τρόπο θα κριθεί η πολιτική συνοχή από τα, τις συνέπειες και τα αποτελέσματά της. Γι' αυτό θα πρέπει να, ε, να, επιδιώξουμε μεγαλύτερη ε, συγκέντρωση των προσπαθειών, προσανατολισμό στα αποτελέσματα και ενίσχυση της ε, πολιτικής συνοχής. Επίσης, οι περιφέρειες θα πρέπει να αποδείξουν τι αποτελέσματα θέλουν να επιτύχουν στην προγραμματική περίοδο γιατί μερικές φορές τα κράτη-μέλη δεν έχουν σαφή στρατηγική και πολιτική ετοιμότητα να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις και μερικές φορές είναι ασαφής και οι στόχοι των κρατών μελών. Τα διαρθρωτικά και παιδιτικά ταμεία θα πρέπει για την περίοδο 2014-2020 να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να ε, τονώσουν την οικονομική τους ε, ανάπτυξη για να διέλθουν από την κρίση. Επίσης θα πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την απασχόληση των νέων. Η ποιότητα εταιρικών σχέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο χάρη στα επενδυτικά ταμεία είναι πολύ σημαντική. Έτσι θα ενισχυθεί η τεχνογνωσία και η εμπειρογνωσία των πολιτικών με τη συμπερίληψη των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Επίσης, στα πλαίσια του νέου Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και την ανάγκη καλύτερης ανταγωνιστικότητα στο παγκόσμιο επίπεδο, τα νέα κράτη-μέλη και μαζί και η Κροατία θα πρέπει να προετοιμαστούν για τις μελλοντικέ επενδύσει και να υιοθετήσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσει, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν ε, τα μέσα του νέου στρατηγικού ταμείου και να μην αφαιρήσουν τα κονδύλια αυτά μόνο τι προηγμένες χώρε. Θα πρέπει και οι νέε χώρε να άρουν τα ε, διάφορα δημοσιονομικά και μάλιστα διοικητικά εμπόδια για να μπορέσουν να προωθήσουν την καινοτομία και να αναπτύξουν και αυτές ε, θύλακες αριστείας. Ευχαριστούμε τους σκιώδης ηγητές, όλος τον κύριο Βαλμίτεμπουργκ. Maar ik wil ook eh, op mijn beurt de rapporteur feliciteren met eh, het voorliggende rapport. Eh, ehm. Ik denk dat het... Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η έκθεση είναι πλήρης, ε, μεστή και πραγματικά επικεντρώνεται στα ουσιώδη. Για τους φιλελεύθερους ε, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις καθυστερείς πληρωμών. Δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική πολιτική συνοχής αν δεν διορθώσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις καθυστερημένες πληρωμές και χαίρομαι που το επισημαίνει ο εισηγητής μας. Σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία αυτή, ιδιαίτερα για τις ε, παραμεθόριες περιοχές και πιστεύω ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και αυτή τη διασυνοριακή διάσταση. Είναι πολύ σημαντικές σχετικές προτάσεις ε, του εισηγητού. Αυτά ως προς σημεία. Υπάρχουν όμως και κάποια αρνητικά. Δεν είναι και πολύ σοβαρά βέβαια, αλλά για να υπάρχει κάποια ισορροπία θα πρέπει να επισημάνουμε και κάποιες αδυναμίες. Ξέρετε ότι είμαστε αρκετά επικριτικοί απέναντι στο επενδυτικό πακέτο του Πρόεδρου Γιούνκερ. Τη μόχλευση τη βλέπουμε στα χαρτιά, αλλά έχουμε μεγάλες αφιβολίες κατά πόσο θα υλοποιηθεί και στην πράξη. Επίσης, το σημείο 14, η έκθεση χαιρετίζει την θεματική συγκέντρωση που συνδυάζει τις επενδύσεις με την αηφόρο ανάπτυξη που δεν αποκλείει κανέναν τη στρατηγική του 2020 και ταυτόχρονα ε, ζητούμε μια ελαστικότητα. Πώς συμβιβάζονται η συγκέντρωση, που είναι πολύ θετική, με την ελαστικότητα που ζητάτε για τις περιφέρειες, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης. Νομίζω ότι αυτή η ελαστικότητα που ζητάτε είναι αντιφατική με την ε, πολυπόθετη θεματική συγκέντρωση. Επίσης ε, λέμε ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις αδυναμίες της οικονομίας για να τις ε, γεφυρώσουμε, να προωθήσουμε την έρευνα, την ανάπτυξη, την ευρυζωνικότητα και να στηρίξουμε τις πιο δύναμες περιοχές της Ευρώπης. Στο σημείο 14 όμως, επαναλαμβάνω, είναι αντιφατικό γιατί από τη μια συγκεντρώνεται και από την άλλη με την ελαστικότητα αφήνεται ένα ξέφραγο αμπέλι για την ε, παρήσυρση πολλών και διαφορετικών θεμάτων, κάτι που μπορεί να υποσκάψει τα θεμέλια της πολιτικής συνοχής και την αποτελεσματικότητά της. Επίσης, μιλήσαμε πριν από λίγο για το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Πρόγραμμα, την Ευρωπαϊκή Ατζέντα. Στο σημείο 25 μιλάτε για την πολιτική για τις πόλεις και δίνεται έμφαση στις μεσαίες και μεγάλες πόλεις. Το επόμενο μας θέμα είναι η ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πόλεις. Ποιες είναι όμως αυτές οι αστικές ζώνες, τα αστικά κέντρα, ποια είναι η σχέση των πόλων με την Ήπεθρο. Γιατί θα πρέπει να στηρίξουμε ταυτόχρονα και τα αστικά κέντρα και την Ήπεθρο. Δεν μπορούμε να δίνουμε την έμφαση μόνο στις πόλεις. Επίσης, θα ήθελα στην έκθεση να μην διαφοροποιήσουμε μεταξύ των μεγάλων πόλων των αστικών κέντρων και των ε, μικρότερης διάστασης. Θα μιλάμε απλώς για... Ευχαριστώ κύριε Βαν Μίλτονμπουργκ. Ο λόγος στον κύριο Αβάνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον ε, εισηγητή για την πρότασή του και θα ήθελα και εγώ να συνεισφέρω ένα-δυο πράγματα. Ε, Έχουμε άλλωστε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να ε, εργαζόμαστε επί του ζητήματος. Όταν αναφέρεστε στην ε, απουσία της εδαφικής διάστασης, συμφωνώ τα κυρίως στη διασυνοριακή συνεργασία, όπως ε, τονίσατε και τώρα, που ουσιαστικά απουσιάζει στην έκτη έκθεση. Εξακολουθεί να είναι κρεμότητα κατά την άποψή μου το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να, δείξει, να αναδείξει τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η διαμεθοριακή συνεργασία, αλλά θα πρέπει εδώ να υπερκεράσουμε κάποιους φραγμούς που επιβάλλουν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ε, το γεγονός ότι προβάλλονται, όπως αναφέρθηκε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στρατηγικές Επενδύσεις, το σχέδιο Juncker, ε, θα πρέπει να μας οδηγήσει να τονίσουμε ακόμα περισσότερο το σχέδιο συνοχής, διότι αυτό θα μπορούσε να ε, ενισχύσει ακόμα περισσότερο την οικονομική κοινωνική διάσταση και τις διαφορές, διότι μπορεί να είναι οι πλουσιότερες περιοχές οι οποίες θα μπορούσαν να υποφοληθούν από τις εγγύησεις του Ταμείου. Ε, επίσης, εάν ο προγραμματισμός δεν μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματα, τότε τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να επιλέξουν το πρόγραμμα Juncker και όχι τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ευρωπαϊκά ε, σχέδια επενδύσεων, που σημαίνει ότι οι διαφορές μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμειγνο, τα διαρθρωτικά ταμεία, τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα που αναφέρθηκε, μας οδηγεί στην ανάγκη να τονίσω ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έτσι όπως είναι παρουσιασμένο. Και επίση, πέραν αυτό τη μακροοικονομική ερωσιμότητα, μα ενδιαφέρουν και διάφοροι όροι μακροοικονομικοί που πιέζουν τι περιφερειακές, ε, περιφέρειες και είναι και ει βάρο τη κοινωνική συνοχή, διότι εμεί χρειαζόμαστε περισσότερε επενδύσει και σταθερότητα και μα ανησυχεί το πώ θα εφαρμοστεί η αρχή τη συνεργασία, δηλαδή οι εταιρικέ σχέσει και οι σχετικέ συμφωνίε, και το αν θα ληφθεί υπόψη στο σχέδιο Juncker από την πρώτη στιγμή τη διαδικασία και η συμβολή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ε, α, επαναλαμβάνω βέβαια ότι αυτό δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις πολιτικές πραγματικότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες φορές ε, το γεγονός ότι τα ίδια τα κράτη επιβάλλουν ένα φίλτρο ε, οδηγεί σε ελλείψεις και η εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχή δεν είναι πάντα η κατάλληλη. Ίσως η έκθεση θα μπορούσε να σταθεί λίγο περισσότερο στην ε, περιβαλλοντική διάσταση της πολιτικής συνοχής, ε, για παράδειγμα τονίζοντας την ανάγκη η βιώσιμη ανάπτυξη να ληφθεί υπόψη ε, όταν θα πρέπει να επιλέξουμε τα ε, κατάλληλα προγράμματα ε, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για το μέλλον θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να πιέζει εντόνω ώστε να έχουμε μια ισχυρή πολιτική συνοχή με επαρκή προπολογισμό και ε, όπως αναφέρθηκε μεγαλύτερε εγγύσει για του νέου και ούτω καθεξή. σα. ευχαριστώ πολύ. Thank you. And Madam Ευχαριστώ θα σπάσω τη ρουτίνα και δεν θα συγχαρώ τον εισηγητή, αλλά θα τον ευχαριστήσω για το σχέδιο έκθεσης. Συμφωνούμε ότι υπάρχουν πολύ καλά σημεία σε αυτή την έκθεση και φυσικά δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά που ήδη έχουν υποθεί. Απλώς να είμαι σαφής προς τις προτεραιότητες μας κατά τη δίδυξη των τροπολογιών. Έχουμε δύο πολύ ξεκάθαρα σημεία. Το πρώτο ήδη είχε αναφερθεί και είναι ότι επιθυμούμε ισχυρότερη έμφαση σε θέματα που αφορούν την πράσινη οικονομία. Οι προτεραιότητες των επενδύσεων που έχουν δοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη και θεωρούμε ότι έτσι δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη Ευρώπη. Αυτό πρέπει λοιπόν να αναφερθεί ε, πιο κατάλληλα και να τονιστεί στην ε, έκθεση ότι δηλαδή η βιώσιμη οικονομία είναι βασικό στατικό της ε, πολιτικής συνοχής και το δεύτερο σημείο αφορά το, την αρχή της εταιρικής σχέσης και του κώδικα διοντολογίας γιατί η πολιτική συνοχή μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν όλοι οι εμπλεκόμενοι ε, και μαζική κοινωνία των πολιτών, τότε μονάχα μπορούν οι επενδύσει να είναι επιτυχημένες. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί επίσης. Και όσον αφορά τώρα το κείμενο, πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν ότι αναφορά στο FC και θεωρώ ότι θα πρέπει και από την πλευρά τη των Περιφερειών να έχουμε έμφαση σε αυτό το σημείο ώστε να τονίσουμε ότι απαιτούμε ότι σε συνδυασμό με την πολιτική συνοχής ότι αυτά τα δύο στοιχεία δεν ε, αντικρούν το ένα το άλλο, ότι μπορούν να συνδυαστούν. Τα θέματα της ευελιξίας. Αν θέλουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι, το ερώτημα που θέτει είναι αν τα κράτη-μέλη θα είναι διαθέσιμα να ευθυγραμμιστούν με τις φιλοδοξίες ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν μιλάμε συγκεκριμένα για βιωσιμότητα και για πράσινη οικονομία. Άρα λοιπόν από την ευρωπαϊκή πλευρά θα πρέπει να πούμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ε, παρόμοιες ε, φιλοδοξίες. Κάνετε λόγο για την κατάχρηση των ε, κονδυλίων. Στην έκθεση θα θέλουμε να γίνει αναφορά, άμεση αναφορά σε θέματα διαφθοράς που έχουν παρατηρηθεί σε κάποια κρατημέλη και σε κάποιες περιφέρειες. Γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε και τη διαφθορά ώστε να είναι η πολιτική συνοχής. Κάνετε αναφορά στην ενεργεία των νέων. Ακόμα δεν υπάρχει σαφή αναφορά στην πρωτοβουλία για την εργασία, την ελληνική απασχόληση. Θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε και αυτό το στοιχείο και να ενισχύσουμε το σημείο αυτό στο οποίο η πολιτική συνοχή ε, υποστηρίζει την ε, εργασία των νέων και καταπολεμά την ανεργία. Και ένα τελευταίο σημείο που αφορά την ε, διοικητική ικανότητα και το χτίσιμο το τίσιμο διοικητική ικανότητα στι τοπικέ αρχέ είναι επίση πολύ σημαντικό ώστε να καταπολεμηθεί η διαφθορά και ώστε η πολιτική συνοχή να γίνει βιώσιμη. Όλο το έγγραφο εστιάζει και στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον της πολιτικής συνοχής. Προσθέτει και νέες διαστάσεις που αφορούν ε, το αποτέλεσμα, την επίδοση. Θεωρούμε ότι και αυτά είναι σημαντικά, αλλά θέλουμε να προσθέσουμε στο θέμα όπου κάνουμε αναφορά στο μέλλον, είναι οι εμπειρίες που έχουμε σύλλεξει κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης, το θέμα της αντοχής, της ανθεκτικότητας. Η πολιτική συνοχή είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε η οικονομία μας να γίνει πιο ανθεκτική και για το μέλλον της πολιτικής συνοχής θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προσθέσουμε και αυτή τη διάσταση. Και κλείνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή για το έργο του και ελπίζω να έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Μαντάμ Ντεμάτο. Κυρία Ντεμάτο. Ε, πάτα Κυρία Νταμάτο, εγώ αντικαθιστώ τη συνάδελφο ε, η οποία είναι αρμόδια για το θέμα γιατί είναι σε άλλη επιτροπή γιατί είναι εισηγήτρια σε κάποια έκθεση. Να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή και θα περάσω σε κάποιες παρατηρήσεις και να μην επαναλάβω αυτά τα οποία είπαν ήδη προλαλήσαντες. Σελίδα 6, παράγραφος 5 ε, της έκθεσης, εδώ αναφέρεται μια ανησυχία για τις καθυστερήσεις της εφαρμογή της προγραμματικής περίοδου 2014-2020 και τα σχετικά προγράμματα. Ε, και εδώ αναφέρεται στην ίδια παράγραφο και η καθυστέρηση κατά 25 δις ευρώ για την περίοδο 2007-2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι και τα δύο θέματα είναι πολύ σημαντικά και δεδομένου ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές επιχειρηματολογίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστές παραγράφους. Οι τοπικές ε, και εθνικές αρχές θα πρέπει να διευκολύνουν το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποβάλλοντας επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία θα συνάδουν με το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημάνουν κάνουμε ότι η καθυστέρηση των προλογών είναι πάρα πολύ σοβαρή, κυρίως mm. γιατί είναι εις αυτών που έχουν κάνει κατάλληλο προγραμματισμό και έχουν κάνει κατάλληλα επιχειρησιακά προγράμματα για την κοινότητα. Δεύτερο, σελίδα 7, παράγραφος 7 για την περίοδο 2014-2020 ίσως η γρήγορη έγκριση θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τονίσουν την ποιότητα των προγραμμάτων, ώστε να αποφύγουμε προγράμματα τα οποία δεν είναι στο ύψος των ε, ε, περιστάσεων, να ε, μην εγκρίνονται απλώς και μόνον για να προλάβουμε τις προθεσμίες. Νομίζω ότι αυτό ισχύει και για την Ιταλία, αλλά και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Έγινε ένας πρώτος γύρος ε, σχολείων από τους και αντισηγητές. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Μπλάνκο Λόπες που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ λακωνικός. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την έκθεσή του και να εκφράσω και κάποιες ε, ανησυχίες που θα τις αποτυπώσω και σε τροπολογίες. Θα υποβάλω εγώ έκθεση για την μακροαρεσιμότητα, ένα ζήτημα που συζητήθηκε εκτερό στο Κοινοβούλιο στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Το θέμα της μακροαρεσιμότητας και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σημαντικό ζήτημα, το ανέφερε και η κυρία Μπρέσο στη δική της παρέμβαση. Θεωρώ ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να εξακολουθεί να αποτελεί την ε, βασική επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα το πω και στην δική μου έκθεση και το διατυπώνω και τώρα. Υπάρχουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των επενδυτικών ταμείων που ίσως υπονομευθούν από τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών εξαιτίας αυτής της μακροαιρεσιμότητας της ε, οικονομικής. Και το να επιφορτήσουμε την πολιτική συνοχής ε, με ευθύνες που είναι άσχετες κανονικά με αυτήν, ουσιαστικά την αποδυναμώνουμε και αποδυναμώνουμε και την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και θα έχουμε αρνητικές ε, συνέπειες και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Γι' αυτό και είμαι κατά της δυνατότητας ε, η μακροοικονομική ερεσιμότητα να αποβεί βάρος ε, του πρωταρχικού στόχου της συνοχής. Θεωρώ ότι η αιρεσιμότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για να αποκλείσουμε τις υπερχρεωμένες περιοχές που εξαιτία της ε, δινής συγκυρίας δεν μπορούν ούτε να επενδύσουν ούτε να προσελκύσουν επενδύσεις εξαιτία τη κακή οικονομική κατάσταση. Σε ό,τι φορά ε, τις παραγράφους 15 και 17 που ακολουθώ αναφέρουν το θέμα, θα υποβάλω τροπολογίε για να διατυπώσω ακριβώ την ανησυχία μου και ουσιαστικά να σας δώσω μία πρόγευση για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει την Επιτροπή επί της δικής μου έκθεσης που αφορά την ε, μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Σας ευχαριστώ. Έξι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Προτείνω να ολοκληρώσουμε έτσι τον κατάλογο των ομιλητών. Άντε και κύριος Πόλτσακ και ο Μαρτζή. Οχτώ συνολικά ομιλητές θα ακούσουμε. Και θα ολοκληρώσουμε τους δικούς μας ομιλ... τη συζήτηση με τους δικούς μας ομιλητές. Ε, κατόπιν θα ακούσουμε τους καλεσμένους μας ε, από την Επιτροπή Περιφερειών ε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ζουλάρ. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Ζουλάρ. Ok, c'est bon. Oui, euh, une collègue a dit qu'il fallait ni féliciter ni remercier. Ε, κάποιος συνάδελφος είπε ότι θα πρέπει ούτε να ευχαριστήσουμε ούτε να συγχαρούμε τον εισηγητή. Κι όμως είναι καλό το έργο του. Είναι χρήσιμο η Επιτροπή μας ε, να χρησιμοποιήσει αυτή την έκθεση ως βάση στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής αιτίας, ε, εμένοντας σε κάποια σημαντικά σημεία της έκθεσης που θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Το πρώτο θέμα αφορά την απλούστευση των διαδικασιών. Αυτό επισημαίνει ο εισηγητής κ. Ντέιτς και η ελάφρυνση των διοικητικών διατυπώσεων για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και για τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά. Δεύτερον, οι περιμερίες, ε, συσσόρευση ανεξόφλητων λογαριασμών, ε, βραδιπορία των επιχειρησιακών προγραμμάτων και πάνω απ' όλα καθυστερημένες πληρωμές. Ε, αυτό το θέμα θα πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μεριμνήσει για τη διόρθωση αυτών των σημείων και των αδυναμιών. Συμπληρωματικότητα επίσης με το επενδυτικό πακέτο του Προέδρου Γιούνκερ. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η συμπληρωματικότητα και η σύνδεση των περιφερειακών πολιτικών με το επενδυτικό πακέτο Juncker. Άλλο σημείο, οι πόλεις. Φυσικά η Επιτροπή μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εδώ όλα μην ξεχνούμε και τις α, μεσαίες πόλεις. Έχουμε πάρα πολλές μεσαίου μεγέθους πόλεις που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντικές λοιπόν αυτές οι παράγραφες της έκθεσης ε, και δίνουν ε, κατευθύνσεις για το έργο της Επιτροπής μας κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής μας θητείας. Γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής. Γιατί είναι κάτι που θα βιώσουν ε, άμεσα οι συμπολίτες μας. Ευχαριστώ. Thank you. And now... Ευχαριστώ, κύριος Πρίος. Ευχαριστώ. Έχω πολλές παρατηρήσεις. Καταρχήν, ε, ε, επενέσατε τα πλεονεκτήματα των ε, κοινωτικών ταμείων, κάτι που δεν βρίσκει πάντα σύμφων στις περιφερειακές αρχές ή όσους ασχολούνται με τα προγράμματα. Για παράδειγμα, την περασμένη Πέμπτη γενιάσαμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα στον Όρπαντε Πάντε Καλέ και ήδη αντλήσαμε κάποια συμπεράσματα. Πολλοί συμμετέχοντες ε, ε, είχαν κακή αντίληψη για τη διαδικασία πρόσβασης σε κοινοτικά κονδύλια. Έκριναν πολύ περίπλοκη αυτή τη διαδικασία. Επίσης ε, δεν αντιλαμβάνονται όλη την ευρωπαϊκή ορολογία που την κρίνουν ιδιαίτερα τεχνοκρατική. Η θεματική συγκέντρωση που σας βρίσκει σύμφωνο και την πρεσβεύετε, δυστυχώς θα αποκλείσει σημαντικά επενδυτικά προγράμματα που θα έχουν, που θα έχουν και σημασία για, την, ε, για τις περιφερειές μας. Τι γίνεται με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό που δεν βρίσκονται ούτε σε θεματική ενότητα, ούτε σε άξονα προτεραιότητας. Νομίζω ότι έτσι θα ε, μπορούσαμε να τα συνδέσουμε με την εδαφική διάσταση. Γιατί είναι κρίμα να αποκλείσουμε με την θεματική συγκέντρωση κάποια σημαντικά προγράμματα. Επίσης, δυσκολίες έχουμε ε, στο να συνδυάσουμε τα κοινοτικά ταμεία με τα ε, προγράμματα των περιοχών και τα, τα, τις τοπικές συμβάσεις. Μιλήσατε για την ε, απορροφητικότητα των κονδυλίων. Οι μηχανισμοί ε, κήρυξη των διαγωνισμών μερικές φορές ε, φέρνουν σε δυσμενή θέση τις μικρές κοινότητες που δεν έχουν τη διοικητική δυνατότητα ούτε είναι ανταγωνιστικές ε, σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα ε, για να υποβάλουν προγράμματα. Χρειάζονται τεχνικής αρρωγής αυτές ε, οι μικρές κοινότητες και δήμοι. Ε, μέλημά σας είναι ο περιορισμός των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών. Αλλά δυστυχώς με τη μορφή που έχουν τα κοινοτικά κονδύλια δυστυχώς τίποτα δεν θα αλλάξουν ως προς τις ανισότητες. Ε, και δυστυχώς ε, μερικές περιφέρειες και κοινότητες αισθάνονται ότι είναι πολύ μακριά από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχή. Και υπάρχει κρίση και με τις πληρωμές. γιατί χρειάζεται μερικές φορές ε, σημαντική οικονομική βάση ε, για να αναλάβει κανείς ένα πρόγραμμα, κάτι που δεν ισχύει για πολλές μικρές ε, κοινότητες και δήμους. Και μάλιστα στη τέλη του 2012 ήταν 38% το ποσοστό πληρωμό, το εκταμίευσης με στόχο το 67%. Με υπερήμερες πληρωμές 25 δις για το 2014. Και μάλιστα η κατάσταση φαίνεται να έχει επιδεινωθεί κάτι που δημιουργεί εύλογες ε, ανησυχίες και στα κράτη-μέλη και στους ε, εταίρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γιατί αυτή η κρίση πληρωμών ουσιαστικά ε, απαξιώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αξιοπιστία της και συγκεντρώνει τις, τις επικρίσεις για αναξιόπιστα και περίπλοκα προγράμματα. Ο κύριος Μπόγκοβιτς είναι ο επόμενος ομιλητής μας. <clears throat> Ευχαριστώ. Και να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στον εισηγητή για την εξαιρετική έκθεση που μας έχει παρουσιάσει. Ήταν ιδιαίτερη χρονική στιγμή στην οποία εκπονέθηκε αυτή η έκθεση. Περικλεί την, ε, το πολιτές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο του 2014 και μετά. βρίσκουν απαντήσει ε, σε ερωτήματα όπως είναι η καθυστέρηση πληρωμών και υποστηρίζω ότι πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα με την καθυστέρηση των πληρωμών. Στο διάρκεια του 2010 2013 αυτό που λείπει είναι μια γενική εικόνα για το τι έχουν πράξει τα κρατη σε αυτό το χρονικό διάστημα. Σε κάποια ε, κράτη-μέλη υπάρχουν ε, μεγάλα προβλήματα όπου το 2014 και 2015 υπάρχουν ε, κονδύλια που έχουν εξαντληθεί και γι' αυτό θα πρέπει να εκφράσουμε την προσδοκία έναντι της Επιτροπής να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό ώστε στα κράτη-μέλη ε, να μην, μένουν, να μην απορροφώνται αυτά τα κονδύλια. Θα μπορούσε και η Επιτροπή με την ε, συνεισφορά της να βοηθήσει την επίλυση του θέματος αυτού τόσο για τα κράτη-μέλη αλλά και για το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή θα ήταν καλό να προφηθούν αυτά τα κονδύλια. Επίσης σημαντικό να υπάρχει μία εκτίμηση ώστε να έχουμε μία βάση για μελλοντικές ε, εργασίες. Κάτι που παρατήρησα στις επισκέψεις της Επιτροπής στα κράτη-μέλη είναι ότι αυτές οι επισκέψεις είχαν φιλική έκβαση και δεν αντικατόπισαν επαρκώς την ε, πραγματική κατάσταση. Το θέμα είναι ότι προκύψαν ε, ε, προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί θα πρέπει να γίνει ε, αναφορά σε αυτά τα θέματα όταν υπάρχουν. Όσον αφορά τις, ε, νέες, ε, τις πολιτικές δημοσιονομικές ε, προπτικές, αναφέρονται και αυτές μέσα στην έκθεση. Θεωρώ ότι είναι πολύ φιλόδοξες. Αυτή είναι μια άλλη προσέγγιση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αποκοινούμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει κάνει μια πρόταση πολύ φιλόδοξη και πολύ ε, ε, πιο ε, επιθετική σε σχέση με την προηγούμενη Επιτροπή. Έχουμε και το πακέτο Γιούγκερ που έχει αναφερθεί ήδη και σε αυτό το πλαίσιο προκύπτει και μια ακόμα ερώτηση, την πρέπει να απαντήσουμε όλοι από κοινού και αυτή η ερώτηση είναι πώς η, κοινωνική, η πολιτική συνοχής θα ενσωματωθεί στο σχέδιο Γιούγκερ, πώς θα ε, αλληλοσυμπληρωθούν αυτές οι δύο πτυχές. Κάνουμε ε, λόγο για ιδιωτικό κεφάλαιο στο πρόγραμμα Juncker αλλά στην πολιτική συνοχής επί της ε, ουσίας κάνουμε λόγο για αύξηση των επενδύσεων στον δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και με αυτά τα σημεία στο πώς χειριζόμαστε το θέμα του σχεδίου Juncker και πώς η πολιτική συνοχή θα λειτουργήσει σε αυτό το χρονικό ε, πλαίσιο ώστε στο μέγιστο βαθμό να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των δύο. Θα πρέπει επίσης να, ε, να προσέξουμε και τα νέα κράτη-μέλη, στο να μην παρουσιαστούν και εκεί προβλήματα λόγω έλλειψης εμπειρίας. τα κράτη-μέλη που προσχώρησαν πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γι' αυτά αποτελεί η πολιτική συνοχή την το, καλύτερο μήνυμα για αυτές τις χώρες και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει σε αυτό το τομέα ε, να καταλάβουμε ότι φέρουμε πολύ μεγάλη υψηλή ευθύνη και να φροντίσουμε στο νέο χρονικό πλαίσιο η πολιτική συνοχή να συνδεθεί με αυτήν την ε, φιλοσοφία. Κύριος Βαμίστερόη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, και από την πλευρά μου θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η ικανοποιητική είναι η έκθεση οποία μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το μέλλον όπως είναι η ενδιάμεση αναθεώρηση. Μας δίνει την ευκαιρία να ονομάσουμε και να αναφέρουμε πολλά θέματα. Η ευελιξία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, παραδείγματο χάρη, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να είμαστε και προσυλλομένοι σε στόχους, θα πρέπει να έχουμε θεματική εστίαση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Όλα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στα σημεία που μας ενδιαφέρουν και δεν θα πρέπει να υπάρχουν αλλαγές. Και αυτό που με εκπλήσει είναι ότι από συνάδελφο που προηγουμένως είπε ότι θα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τα πάντα, ε, γήπεδα γκολφ και τα λοιπά. Προσθέμενη αξία μας είναι ότι έχουμε και τη δυνατότητα να επιλέγουμε. Να ε, ενισχύσουμε την εργασία των νέων, Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σκορπίσουμε κονδύλια σε όλη την Ευρώπη βέβαια. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη. Αυτό είναι που μας αφορά. Θα πρέπει να μείνουμε ευθυγραμμισμένοι προς αυτό. Ναι, βέβαια, από τη μία πλευρά υπάρχει ευελιξία στο πλαίσιο των 7 ετών, αλλά θα πρέπει να έχουμε έναν ρυθμό και σε δύο χρόνια να εφαρμόσουμε επιχειρησιακά σχέδια. Θα μπορούσα να πω λοιπόν τη νέα επιτροπή. Έχει όντως μια νέα προσέγγιση. Θέλει καλύτερη νομοθεσία. Όντως σε αυτό το σημείο μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά πράγματα και αυτό θα το ενισχύσει πολύ και μια ενδιάμεση αναθεώρηση. Θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να προσαρμοστεί σε αυτό και να στηρίξει το ρόλο του και η κυρία Μπρέστο το ανέφερε επίσης. Το δεύτερο στοιχείο που μου λείπει στην έκτη έκθεση για τη συνοχή είναι αυτή η συνέργεια ανάμεσα στα ταμεία. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την ύπεθρο, με την ενέργεια, με τον ορίζοντα 20, 2020 κτλ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τα ταμεία. Είναι τα ταμεία και θα πρέπει να φροντίσουμε ε, το 30% των δηλίων να ε, <coughs> επενδύονται στις υποδομές και σε αυτό το επίπεδο μπορεί να υπάρξει συνέργεια και υπάρχουν και συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μονομένες ε, νομοθεσίες και τα οποία μπορούν να προσφέρουν νέες δυνατότητες για περιοχές, περιφέρειες και να συνδυαστούν με άλλα τα μία κονδύλια που ειδικεύονται σε συγκεκριμένα ε, πράγματα. Να δημιουργηθούν αυτοί οι σύνδεσμοι ανάμεσα στα διαφορετικά χρηματοδοτικά ε, μέσα. Να προωθηθούν επίσης μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά μπορούν να προσθεθούν ε, ε, στην έκθεση. Λείπουν από την έκθεση και ε, όσον αφορά την εδαφικότητα, Ε, υπάρχει αυτή η μέση διάταξη ε, για τις επικράτειες η οποία προβλέπεται και από τη συνθήκη της Λισαβόνας, αυτός ο τρίτος ε, στόχος να υπάρχει κοινωνική, οικονομική και δαφική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση αναφέρεται ότι θα πρέπει το 2015 να γίνει αξιολόγηση. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί λόγοι για να γίνει όντως αυτό. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο το, στα του 2015. Όποτε θα γίνει και η εξολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης γίνεται αναφορά και στην, στο ρόλο των πόλεων στο θέμα της εδαφικής ε, συνοχής. Κομοπόλεις, οι μεσαίες μεγάλες πόλεις όλα αυτά θα μπορούσαν, θα μπορούσαν να συνδεθούν με συγκεκριμένου στόχους. Πολλοί δεν είναι ικανοποιημένοι με το θέμα αυτό και με την εδαφική ημερήσια διάταξη. Όταν κάνουμε λόγο για συνεργασία, σε αυτά έχουμε μείνει πίσω. Και αν τα συγκρίνουμε όλα αυτά με την ε, παρούσα έκθεση για τη συνοχή, έχουμε την αίσθηση ότι κάτι λείπει και ότι δεν συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά. Θα επανέλθουμε βέβαια στο θέμα του σχεδίου Juncker, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία που θα μπορούσαν να τονιστούν περισσότερο στην έκθεση του κυρίου, του κυρίου Deutsch. Ευχαριστώ. Κυρία Μαλέτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το συνάδελφό μας ε, Τάματς για αυτή την ε, άρτια ε, έκθεση. Πρόκειται για μια έκθεση ιδιαίτερη σημασία και για μας και για την Επιτροπή μας και θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία. Πρώτον, οι προσπάθειές μας να υπάρχει ανάπτυξη, ε, η πολιτική συνοχής να είναι αναπτυξιακή ε, πολιτική και δεύτερον είναι το θέμα της καθυστέρησης εφαρμογής ε, για το διάστημα 2014 έως το 2020. Όσον αφορά το πρώτο, θεωρώ ότι θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να υπάρχουν περισσότερα προγράμματα τα οποία θα είναι αφιερωμένα στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ε, προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης, όχι μόνο προγράμματα υποδομών, αλλά και τέτοιου ίδιους προγράμματα και αυτό φυσικά είναι και ο ρόλος μας, ε, να ε, προασπίσουμε αυτά τα προγράμματα στις χώρες μας, διότι... Υπάρχει ένα νέο ταμείο για στρατηγικές επενδύσεις, ένα νέο σχέδιο επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι οι τρεις σημαντικοί πυλώνες σε αυτό το σχέδιο είναι η χρηματοδότηση ως μορφή επένδυσης, ε, όπως το έχουμε και στην πολιτική συνοχή, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, αλλά επίσης και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ε, αυτός είναι ο δεύτερος πυλώνας και ο τρίτος πυλώνας είναι ε, καλά προετοιμασμένα και διαρθρωμένα προγράμματα τα οποία συνάδουν και με την πολιτική ανάπτυξη των χωρών. Και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει ε, να το τονίζουμε όταν συζητούμε την πολιτική συνοχή και όταν χρησιμοποιούμε τις ε, μορφές χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό θα πρέπει να προσπαθούμε να εναρμονίσουμε τις νέε προσπάθειες τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αυτό το νέο επενδυτικό σχέδιο και τις προσπάθειες που κάνουμε στην πολιτική συνοχή. Θα πρέπει κάπως αυτά να εναρμονιστούν και να κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση. Δεύτερον, όσον αφορά την καθυστέρηση στην εφαρμογή, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 80% εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλά ταυτόχρονα βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος των δημοσιονομικών προοπτικών και ήδη ε, ε υστερούν αρκετά στα κράτη-μέλη όσον αφορά την, ε, τις ε, ε, τους εκ των, όρους ε, που βασίζονται στους όρους αυτούς, ε, στρατηγικά έγγραφα, ανάλυση που πρέπει να έχουν προετοιμαστεί ήδη στα κράτη-μέλη. Και επίσης θα πρέπει να ολοκληρώσουν το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για το 2014-2020 και ε, τη διαδικασία πιστοποίησης των δομών. Βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος ε, των προοπτικών. Επομένως, η εφαρμογή σίγουρα έχει καθυστερήσει και βρίσκεται σε κίνδυνο. Υπάρχει ο κανόνας του νησιν 3, αλλά ε, πλέον δεν είναι νησιν 3, είναι νησιν 2 και ακόμα και λιγότερο και επομένως θα πρέπει να δούμε τι μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν προκειμένου να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την εφαρμογή και να μην υπάρχει απώλεια ε, δεσμεύσεων ε, ε, υποχρεώσεων για το 2017. Ευχαριστώ. Τώρα θα μιλήσει υποφαινόμενη και θα μιλήσω βουλγαρικά. Διότι θα λάβω το λόγο προκειμένου να σχολιάσω την γνωμοδότηση. Να ευχαριστήσω το συντάκτη της γνωμοδότησης για την πολύ καλή δουλειά του και την επικοδομητική του στάση επί του ζητήματος και τα όσα μας παρουσιάζει στην γνωμοδότηση. Ε, όπως ακούσαμε από τις συναδέλφους, τα περισσότερα πόσα λέει ε, αντανακλούν και τη δική μας την άποψη για την έκτη έκθεση συνοχής. Θα ήθελα να υποστηρίξω πλήρως το γεγονός ότι ε, στέκεται στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής εν καιρό κρίσης και τις συνέπειες ε, για την πολιτική συνοχής λόγω της κρίσης και το πώς η πολιτική συνοχή βοήθησε να μετριαστούν οι συνέπειες της κρίσης σε πολλές ε, χώρες μέλη. Η έκτη έκθεση καταδεικνύει ότι κάποια από τα μέτρα στις επενδύσεις ε, ε, για την πολιτική συνοχή υπερβαίνουν το 60% των εθνικών επενδύσεων συνολικά. Και είναι πολύ σημαντικό να σχολιάσουμε το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής ε, ε, έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να ενισχύσει το επίπεδο επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζω την προσέγγιση που ε, έχει επιλέξει ο εισηγητής ε, ζητά συμπληρωματικότητα και συνέργεια μεταξύ της πολιτικής αυτής και των άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ως προς τις συνέργειες και, την και τη συμπληρωματικότητα όχι μόνο την ανάγκη για τις στρατηγικές επενδύσεις, ε, το λεγόμενο σχέδιο Juncker δηλαδή, αλλά να υπάρχει συμπληρωματικότητα με όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι τελικώς όλες οι πολιτικές ε, εφαρμόζονται εφαρμόζονται εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Επομένως, το αποτέλεσμα μπορεί να έχει πολλαπλασιαστική επίδραση και αν δεν υπάρχει συμπληρωματικότητα και συντονισμός των στόχων μας, τότε θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι ε, μετριότερο το αναμενόμενο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το οποίο τονίζεται στην έκθεση και πιο συγκεκριμένα το γεγονός ότι δεν δίνεται ε, αρκετή έμφαση στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής συνοχής, διότι είναι κάτι το οποίο γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις άλλες ε, πολιτικές και η εδαφική διάσταση μας δίνει και μια εικόνα των συγκεκριμένων εδαφικών αναγκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και ακριβώς υποστηρίζω την προσέγγιση ε, να αναζητήσουμε συγκεκριμένους στόχους για κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο της έκθεσης ε, που έχει τονιστεί ιδιαιτέρως. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε και τη στρατηγική σημασία των ε, πόλεων μεσαίου μεγέθους, όχι τόσο των μεγάλων πόλεων. Αν δούμε την πιο πρόσφατη μελέτη της Epson, που μας δίνει και ένα μοντέλο ε, για την Ευρωπαϊκή Επικράτεια μέχρι το 2050 ε, διαπιστώνουμε ότι οι μεσαίου μεγέθους πόλεις θα διαδραματίσουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εδώ στην έκτη έκθεση συνοχής να τονίσουμε το ρόλο αυτής της εξέλιξης. Σίγουρα θα είναι όλο και πιο σημαντικά τα διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα και θα πρέπει να τα τονίσουμε και αυτά στην έκθεσή μας και τη σημασία τους για την πολιτική συνοχής επίσης. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό με το σχέδιο Γίνκερ αλλά και με άλλες πολιτικές. Και με αυτό ολοκλήρωσα και τώρα να δώσω ε, το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια στοιχεία αυτής της έκθεσης. Ε, θα, καταρχάς να συγχαρώ το συντάκτη της γνωμοδότησης γιατί αυτό το οποίο του ανατέθηκε ήταν ε, ένα ευρύτερο πεδίο και νομίζω ότι το αποτέλεσμα αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τις εργασίες μας. Οι σκιώδεις συντάκτες... Ε, ε, παρουσίασαν και μία σειρά από τροπολογίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την έκθεση. Να σας πω ότι οι καθυστερήσεις καταρχάς αποτελούν ε, μείζον πρόβλημα και αυτό ε, αναφέρεται δεόντως στην έκθεση. θεωρώ ότι ούτως ή άλλως σταθήκαμε σε αυτό επαρκώς, επομένως δεν θα ήθελα να πω εγώ περισσότερο. Θα ήθελα να τονίσω όμως λίγο περισσότερο το θέμα της απασχόλησης ο συντάκτης τονίζει το θέμα της απασχόλησης των νέων. Και κατά την άποψή μου δεν πρόκειται μόνο για ένα κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, αλλά πρόκειται και για ένα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται ε, και ε, με ένα βαθμό κινδύνου. Η ανεργία των νέων είναι γόνιμο έδαφος ε, για ε, τον εξτρομισμό, αποτελεί γόνιμο έδαφος για παθογένειες όπως η τρομοκρατία, η οποία εκδηλώνεται ή εκδηλώθηκε ήδη και στο Παρίσι και στην Κοπενχάγη και σε άλλες πόλεις. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κάποια στατιστικά στοιχεία της ανεργίας των νέων κυρίως ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Ε, βέβαια δεν επαφίεται στον ε, συντάκτη της νομοδότησης να το συμπεριλάβει αυτό στην έκθεση. Θα μπορούσαμε να το προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα και θεωρώ ότι αυτό θα μας επιτρέψει να αντιληφθούμε λίγο καλύτερα και την ε, κοινωνική συνοχή και τις απαραίτητες επενδύσεις για την απασχόληση και την, και την ανάπτυξη. Δεύτερον, στην ε, γνωμοδότηση αναφέρεται ότι οι επενδύσεις ε, πέρασαν από τις υποδομές ε, προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τις πολιτικές απασχόλησης, τις πολιτικές καινοτομίας και ούτω καθεξής. Αυτή η μεταφορά όντως έγινε και εδώ θα ήθελα να τονίσω και πόσο σημαντική είναι η συνέργεια. Ο κύριος Βανίστερλοϊ αναφέρθηκε ήδη στο θέμα αυτό στην παρέμβασή του και θεωρώ ότι οι συνέργειες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ε, στην ανάπτυξη των μικρών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, σε καινοτομία αλλά και σε επενδύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν και σε επίπεδο υποδομών. Τονίζω λοιπόν πόσο σημαντικές είναι αυτές οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα. Και μια τελευταία παρατήρηση για το σημείο 16 της έκθεσης. Στο σημείο 16 τονίζεται η ευθύνη του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εποπτεία. Πρόκειται για το άρθρο 23, το οποίο πλέον πρέπει να εφαρμοστεί και να υπάρξει και ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα αξιολογήσει κατά πόσον εφαρμόζεται το άρθρο αυτό. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, διότι η αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ ισχυρέ. Πρόκειται για αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εάν το μέσο αυτό χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κανόνες εφαρμογής του συγκεκριμένου μέσου θα πρέπει να είναι ε, καθόλου ακριβείς. Ο κύριος ε, Λόπεθ, ε, ο αρμόδιος εισηγητής, θα εξετάσει το σημείο αυτό. Εγώ θα είμαι σκιώδης εισηγητής από πλευράς ΕΛΚ και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, τονίσουμε την ακρίβεια και την προβλεψιμότητα αυτής της διαδικασίας που σχετίζεται με το άρθρο 23. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητή στη συζήτηση αυτή, ο κύριος Όμερσελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το πολύ αξιόλογο έργο του ε, και ως προς τη διάγνωση και τις διαπιστώσεις που έκανε της κατάστασης και ως προς τις προοπτικές, ιδιαίτερα για την περίοδο μετά το 2020. Δεν πρόκειται να επαναλάβω όσα ήδη ακούσαμε. Θα ήθελα να σταθώ σε λίγα μόνο σημεία. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο Juncker, το επενδυτικό πακέτο όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι, είμαστε υπέρ αυτού του σχεδίου Juncker. Ελοχεύει όμως ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος. Το κατά πόσο θα φτάσει στις αναγγελίες και στις υποσχέσεις, τα 315 δισεκατομμύρια δηλαδή των επενδύσεων. Πολύ φοβόμαστε ότι αυτό το σχέδιο τελικά θα αποσταθεροποιήσει όλο το μέχρι τώρα οικοδόμημα της συνοχής φοβόμαστε μήπως ε, τελικά αυτό το επενδυτικό σχέδιο επιδεινώσει τις ε, περιφερειακές ανισότητες, γιατί 300 δισεκατομμύρια ευρώ είναι περίπου ολόκληρος ο προϋπολογισμός της περιφερειακής πολιτικής. και περίπου ο προϋπολογισμός της κοινή γεωργικής πολιτικής. Έχω κάποιες αφιβολίες λοιπόν για το κατά πόσο θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτά τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Θεωρητικά όμως αν έχει κανείς 300 ε, δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στις περιφέρειες δημιουργούνται τεράστιες ευκαιρίες αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη κίνδυνη να αμφισβητηθεί το μέχρι τώρα επίτευγμά μας ε, στην πολιτική της συνοχής. Η ίδια η συνοχή δηλαδή να υπονομευθεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται αυτό το σχέδιο Γιούνκερ γιατί βρισκόμαστε στην αρχή της νομοθετικής διαδικασίας και η Επιτροπή έχει υποβάλει διάφορες προτάσεις. Γνωρίζουμε όμως ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και ότι αυτή τη στιγμή ο Αντιπρόεδρος ε, ε, κατά Κατάινεν επεξεργάζεται αυτές τις προτάσεις. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να επανέλθουμε σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση και να στηρίξουμε, θα το συζητήσουμε βέβαια και με τους συντονιστές, ε, κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες της δικής μας Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, ίσως αποκινούμε την Επιτροπή Περιφερειών, για να φροντίσουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Αντιπρόεδρος ε, Κατάινεν να δεσμευτούν ε, και να σεβαστούν τους πρωταρχικούς στόχους της περιφερειακής πολιτικής. Τώρα, για τις προοπτικές μετά το 2020. Σίγουρα από τώρα θα πρέπει ε, να αρχίσουμε τις εργασίες ε, για το σχέδιο προγραμματισμού μετά το 2020 και ε, είμαι υπέρ του σημείου Β που αναφέρεται στη σελίδα 5 γιατί ε, αδιαλείπτω στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία τονίζαμε την ανάγκη η πολιτική συνοχής να μην επικεντρωθεί μόνο στις, ε, στους στόχους στρατηγικής 2020 αμελώντας τους στόχους της συνοχής, της σύγκλησης αλλά και της αλληλεγγύης όπως είπε η κυρία Μπρέσο. Γιατί η περιφερειακή πολιτική ίσως είναι η μοναδική ε, μείζον πολιτική αλληλεγγύης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό η Επιτροπή μας ε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πολιτική αυτή. Επίσης, το συνέ... η συνέργεια μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Πολύ σημαντικό και συμμερίζομαι απόλυτα αυτά που είπε ο συνάδελφος ε, Λάμπερτ Βανίλ Αν θέλουμε συγκεκριμένη και αυτή προσέγγιση, χρειαζόμαστε και συνέργεια πολύ συχνά στις επαφές που έχω με τις γαλλικές περιφέρειες διαπιστώνω ότι έχουν επίγνωση για το τι κονδύλοι υπάρχουν ε, ε, για την πολιτική συνοχή, αλλά δεν γνωρίζουν τα υπόλοιπα διαρθρωτικά ταμεία. Τα ταμεία, για παράδειγμα, και τα κονδύλια που τον ορίζοντα 2020, αλλά και κονδύλια της κοινή ιωρικής πολιτικής, γιατί και εκεί θα μπορούσαμε να ενεργοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε κάποια κονδύλια για την έρευνα στην κοινή γεωρική πολιτική. Μάλιστα, πρόκειται για κονδύλια που είναι αρκετά ταψιλή, αλλά άγνωστα στι περιφερειακέ αρχέ. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ενημέρωση, πληροφόρηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Με, τις, με συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για να κατατοπιστούν οι περιφέρειες για τις δυνατότητες που έχουν και τα κονδύλια που μπορούν να αξιοποιήσουν. Επίσης, ε, μιλούμε για την αστική ατζέντα, το αστικό θεματολόγιο. Σήμερα δεν μπορούμε να ε, υιοθετήσουμε μια σφαιρική προσέγγιση, γιατί έχουν διαφορετικά προβλήματα οι πόλεις και ιδιαίτερα τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι μεσαίου μεγέθους πόλεις. Οπότε δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι εξαιτία των μεγάλων διαφορών που υπάρχουν. Έχουμε κάποιες περιφέρειες ε, και πόλεις, αστικά κέντρα που βρίσκονται στην καρδιά της Ευρώπης, μεν, γεωγραφικά, αλλά δυστυχώς ε, βρίσκονται στην περιφέρεια σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Γιατί η συγκέντρωση ε, της ανάπτυξης γίνεται στις μεγάλες μετροπόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα να, να περιθωριοποιούνται κάπως οι μεσαίες πόλεις. Και τέλος, για τις πληρωμές. Επισημάναμε τα προβλήματα, αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκε αηφόρος λύση. Και διατρέχουμε τον κίνδυνο και πάλι το 2017 ή 2018 να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό ίσως θα πρέπει κάπως ε, να επιδείξουμε προνοητικότητα και από εκείνο με την Επιτροπή Προϋπολογισμών να υποβάλουμε προτάσεις για να μην βρεθούμε μετά από λίγα χρόνια στα ίδια προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριο Άλμπερτ Μπορ. Θα κάνει μια σύντομη παρέμβαση εκπροσωπώντας την Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι ο πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών. Ε, πρόεδρος του Συμβουλίου της πόλης του Birmingham και θα μας παρουσιάσει την τοποθέτηση της Επιτροπής των Περιφερειών. Ο λόγος ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, εισηγητή και συνάδελφοι που δίνουν την ευκαιρία να σχολιάσω την έκτη έκθεση πολιτική συνοχή. Η πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από του πυλώνε πάνω στου οποίου ε, στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολιτική που είναι θεμελιώδη για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και επιπλέον είναι μια πολιτική που είναι απαραίτητη για να ε, βοηθήσει την Ευρώπη στην οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική κρίση την οποία διανύουμε μας έχει καταδείξει ότι η ευρωπαϊκή Πόρνη είναι αναγκαία για να διατηρήσουμε το ύψος των επενδύσεων στις ε, περιφέρειες. Πρέπει να δράξουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και να υποστηρίξουμε μια πιο ισχυρή πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολύ κάνατε αναφορά ε, στον αντίκτυπο που θα έχει το σχέδιο του Juncker οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο θα ενισχύσει τη σημασία της πολιτικής συνοχής τα επόμενα χρόνια. Οι βασικές συστάσεις που κάνει στην γνωμοδότηση της Επιτροπή ε, των Περιφερειών για την έκτη έκθεση συνοχής συμπεριλαμβάνει κάποιες, ε, ε, κάποια θέματα που αφορούν στο μέλλον της πολιτικής συνοχής. Θέλουμε μια οικονομικά πιο στεναρή πολιτική συνοχή, η οποία θα διαθέτει περισσότερου πόρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση, θέλουμε μια πολιτική η οποία θα αφορά όλε τι ε, διοικητικέ αρχέ, από τι Βρυξέλλε μέχρι τη μικρότερη διοικητική αρχή και που θα συνεισφέρει στην, ε, στον μοτερνισμό αυτών των διοικητικών αρχών, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στον ιδιωτικό τομέα και να αποτελέσουν ε, όχι εμπόδιο, αλλά έναν παράγοντα ανάπτυξη Επίσης, να ενημερώνονται καλύτερα οι πολίτες ε, για τα αποτέλεσμα που μπορεί να επιφέρει. Να εμπλέκονται περισσότερο στον ε, διάλογο, επίσης ε, για την πολιτική συνοχή. Σε σχέση με όλα αυτά, επομένως, θα ήθελα να καλωσορίσω την εξαιρετική συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών, το 5 και το τροπίζει ε, πολύ επιτυχώς ε, τον το διαθεσμικό ε, διάλογο για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της πολιτικής συνοχής στις περιφέρειες. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ντότζ, τον εισηγητή, για την εξαιρετική του εργασία και την προθυμία του να ακούσει τις συστάσεις που παρουσιάσαμε ως Επιτροπή Περιφερειών. επιπλέον να υπογραμμίσω ε, κάποιες προτάσεις από τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Κατά πρώτον, είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση που γίνεται στην ε, έκθεση για την πολυπεδη διακυβέρνηση ως μια αποτελεσματική δομή ώστε να ανταποκριθούν, να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων τοπικές αρχές είναι υπεύθυνε για τις ε, τοπικές επενδύσεις, όπως τόνισε ο εισηγητής. Επομένως είναι σημαντικό η πολιτική συνοχή να παίξει, ε, να σε σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των δημόσιων αρχών ε, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πρωτίστως, ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ποιότητας στο κοινό. Επίσης, συμμεριζόμαστε τις ε, ανησυχίες που έχετε για την καθυστέρηση ε, της εφαρμογής ε, πολιτικών συνοχής για το 2014, 2014 και το 2015 και για την εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων. Όλα αυτά πλήττουν την αξιοπιστία της πολιτικής συνοχής, συνοχής και την εφαρμογή των διαστοτικών ε, κονδυλίων, την απορρόφηση. Θα πρέπει να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να προσπαθήσουμε να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα καταπολεμώντας ε, τη διαφθορά. Επίσης, ε, θα μειωθούν και τα λάθη αν εξορθολογιστεί η εφαρμογή. Αυτό που τονίζει το σχέδιο έκθεση είναι να υπάρχει συμμόρφωση με τις διατάξεις σε σχέση με την εδαφική συνοχή. Επίσης, ε, καλείται η Επιτροπή να δώσει προσοχή στις ευάλωτες περιοχές όσον αφορά ε, τη δημογραφική εφαρμογή της ε, πολιτικής συνοχής επιπλέον. Να αναφερθώ σε κάποια σημεία τα οποία δεν αναφέρονται στην έκθεση, στο σχέδιο έκθεσης και τα οποία ενδιαφέρουν όμως πολύ την Επιτροπή των Περιφερειών. Θέλουμε να επαναλάβουμε το αίτημά μας, οι δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών, τοπικών και περιφερειακών αρχών να αποτελέσουν ε, μέρος, ε, μέρος ως μέσο ε, χρηματοδότησης να μην συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο ανάπτυξης. Θα θέλουμε να αναλογιστούμε βαθύτερα το ρόλο της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Επενδυτικού Ταμείου και για τις αρμοδιότητές τους. Ίσως δεν θα είναι, θα κατάλληλο να εφαρμοστούν, ε, να δοθούν κονδυλία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ε, εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Επίσης, επαναλάβαμε τις ανησυχίες μας για τον κίνδυνο που υπάρχει στα θέματα της μακροαιρεσιμότητας και για το γεγονό ότι υποσκάπτονται τα προγράμματα επενδύσεων από τις μακροοικονομικές ε, προοπτικές. Επίσης θα θέλουμε να επιμείνουμε ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από το ΑΕΠ και να δούμε περισσότερο τις ε, περιφερειακές προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε σε πιο συγκεκριμένο ε, επίπεδο. Το να επαφιόμαστε στο ΑΕΠ των περιφερειών έχει μειονεκτήματα τα οποία αποσκάπτουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής ε, συνοχής και για την ε, πίστοση κονδυλίων ε, από το Ταμείο Στρατηγικής Στρατηγικών Επενδύσεων. Οι περικοπές επίσης έχουν εμποδίσει τομείς που μπορούσαν να αποφέρουν ανάπτυξη. Γι' αυτό θα πρέπει να αξιολογήσουμε με προσοχή και να λάβουμε υπόψη την, ε, τον αντίκτυπο που έχουμε στην ανάπτυξη και στην απασχόληση ε, μέσω της ε, αναστολής των πληρωμών. Αυτά αναφέρονται στο σημείο 16 της εκθεσής σας. Και τέλος, θα θέλαμε να υπάρχει ένα Συμβούλιο Πολιτικής Συνοχής Αυτό θα μπορούσε να ε, αναδείξει το προφίλ ε, της πολιτικής συνοχής και να εξασφαλίσει έναν ε, πολιτικό διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συμμετάσχει ενεργά στις διάφορες πολιτικές συζητήσεις με θέμα αυτή την δομή, ώστε να διασφαλίσει την πλήρη συνεξιτήμηση των απόψεων των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Αυτές είναι οι προτάσεις από την Επιτροπή των Περιφερειών και θα μπορούσαν να συντηθούν περαιτέρω από την Επιτροπή για την Περιφερειακή Ανάπτυξη να ληφθούν υπόψη τελική, στο τελικό σχέδιο έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και να δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής <coughs> Επιτροπής, τον κύριο Ρούλς Ντέξτρα. Σας ευχαριστώ. Προφέρετε και πολύ ωραία το επώνυμό μου. Είμαι... Ε, εγώ συνέταξα την έκτη έκθεση συνοχής ε, από τη Γενική Διεύθυνση Ρίτζο. Βέβαια είναι αδύνατο να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα και τις απορίες ε, που προέκυψε αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα επικεντρωθώ στα ουσιώδη και θα σας ενημερώσω για τις θέσεις και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχήν να υπογραμμίσω ότι Εστενιζόμαστε τις, τους προβληματισμούς για τις καθυστερημένες πληρωμές και θα φροντίσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Βέβαια, δεν είμαστε οι μόνοι αρμόδιοι για το πρόβλημα αυτό. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία του Συμβουλίου και των κρατών μελών για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα. Τώρα, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα προγράμματα ώστε να επιτρέψουμε σωστή και απρόσκοπτη εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και στη νέα περίοδο προγραμματισμού. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σημείο που έθιξε ο εισηγητής ο κύριος Ντόιτς, για τη διαφορά δηλαδή μεταξύ της Ευρώπης του ορίζοντα 2020 και της υποχρέωσης της, ηθίκη να, της υποχρέωσης ηθίκης να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Δεν βλέπουμε αντίφαση μεταξύ των δύο στόχων, γιατί η κατανομή των κονδυλίων ευνοεί κυρίως τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Και θα το διαπιστώσετε αυτό και στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού. Και δεν υπάρχει διαφορά σχέση με τη μέχρι τώρα μας δέσμευση να στηρίξουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Και πιστεύουμε ότι μετά την διέξοδο και από την κρίση θα μειωθούν οι ανισότητες. Τώρα σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα προαπαιτούμενα για τους θεματικούς στόχους και εκεί λαμβάνουμε υπόψη την ανάπτυξη των περιοχών. Οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ε, απολαμβάνουν μεγαλύτερη ελαστικότητα και ευελιξία. Και νομίζω ότι είναι, ε, δεν είναι περίεργο να ε, σκεφτόμαστε τι θα γίνει με την επόμενη προγραμματική περίοδο όσο ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει την προηγούμενη αλλά και η επόμενη 7η πρόταση, ε, έκθεση συνοχής του 2017 θα περιλαμβάνει προτάσεις για, το επόμενο, για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Και προς τα τέλη του 2017 θα υποβάλουμε και τη νέα πρόταση για τη νέα περίοδο. Νομίζω ότι έτσι θα καταφέρουμε να προετοιμαστούμε άρτια για την ε, συζήτηση. Σε ό,τι αφορά την ε, περιφερειακή συνεργασία και τη διασυνοριακή συνεργασία, σημειώνουμε την πρότασή σας ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για τις παραμεθόριες περιοχές, ούτε ποσοτικά αξιόπιστα, ούτε και ποιοτικά. Και προσπαθούμε με τους εταίρους μας ε, να βελτιώσουμε τις μετρήσεις μας και να διαπιστώσουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές και ευελπιστούμε ότι στην 7η έκθεση συνοχής ε, θα παρουσιάσουμε βελτιώσεις στο θέμα αυτό με συγκεκριμένα από τα παραδείγματα. Σε ό,τι αφορά το στόχο απλούστευσης, η Επίτροπος Κρέτσου έχει δεσμευτεί για να βελτιώσει την εφαρμογή της πολιτικής ε, επιφέροντας ε, απλουστεύσεις. Σε ό,τι αφορά τη διοικητική ικανότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σίγουρα αισθενιζόμαστε την ανησυχία σας για μείωση της γραφειοκρατίας και περιορισμό του γραφειοκρατικού άχθους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα να δούμε τους παγκόσμιους γνώμονες και τους κριτήρια αναφοράς ε, της Παγκόσμιας Τράπεζας, ε, λίγες χώρες ε, είναι κάτω από το βασικό δίκτυο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Θα συνεργαστούμε με αυτές για να βελτιωθούν και στη συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποια περιφερειακά στοιχεία για το easy doing business, για τη βελτίωση αυτής της πρόσβασης. Σε ό,τι αφορά την μακροοικονομική αιρεσιμότητα, σχεδόν ταυτόχρονα με την έκτη έκθεση συνοχής, ε, δημοσιεύσαμε και ανακοίνωση για τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Και θα είμαστε ιδιαίτερα διαφανείς ε, για το πότε και πώς θα εφαρμόσουμε αυτόν τον όρο. Φυσικά ένα σκέλος είναι υποχρεωτικό μετά την καταστρατήγηση της διαδικασίας για το υπερβολικό χρέος θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η δική μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Και αυ... τώρα για το κατά πόσο αυτός ο πυλώνας θα, θα δημιουργήσει πρόβλημα, όχι, είναι μια αυτόματη διαδικασία που κινητοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τον κανονισμό. Για τη συνέργεια μεταξύ των ταμείων, σημαντικό αυτό το θέμα, και η ίδια η έκτη έκθεση συνοχής ε, δεν αναφέρεται διεξοδικά στο θέμα αυτό, αλλά οι προετοιμασίες για τα τρέχοντα προγράμματα δείχνουν ότι σε κάποια προγράμματα έχουμε αυτή τη διάσταση της συνέργειας των πολλών ταμείων. Για παράδειγμα, το Γεωργικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Περιφερειακό Ταμείο εξετάζουν για το πώς ε, θα χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα προγράμματα σε περιοχές ώστε να έχουμε σαφή κατανομή των ε, έργου, του έργου και να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Βέβαια και αυτό το θέμα επιδέχεται βελτιώσεις. Πολλά σχόλια άκουσα για την ισορροπία μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων των μεσαίων μεγέθους πόλεων και της υπαίθρου. Το ζήτημα αυτό το πραγματευτήκαμε και στην έκτη έκθεση συνοχής και θα το αναπτύξουμε περαιτέρω. Στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, πολλές χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης ε, έχουν πια εξίσου ανεπτυγμένες πρωτεύουσες και νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε και τις μεσαίες πόλεις. Βέβαια, ανάλογα με το που διαμένει κανείς, ε, μπορεί να έχει παράπονα αλλά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού έχουμε βελτίωση ε, γιατί χρηματοδοτούμε εξίσου και τις μεσαίες, περι... πόλεις σε σχέση με τις πρωτεύουσε. Και το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής ε, ενίσχυσαν πολύ περισσότερο την Ήπεθρο στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού σε σχέση με, τις, με τα αστικά κέντρα. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν είχαμε μια προκατάληψη βάρος της Ήπεθρου σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχής. Και μην ξεχνάτε ότι και σε αυτή και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα διαθέσουμε μέσω του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης δαψιλή κονδύλια και για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Τώρα, για τρεις περιοχές είχαμε για την περίοδο 2013 ε, χρηματοδοτήσεις με βάση το νήσι, στις περιοχές ΝΑΤΣ και θα δούμε ε, ποιες είναι οι κατανομές των κονδυλίων μεταξύ των τριών ε, επιπέδων. Βέβαια, μπορεί να ε, έχετε αφιβολίες για την ενίσχυση, για την ένταση της ε, ενίσχυσης, αλλά πιστεύω ότι με τη μελέτη που θα κάνουμε θα δούμε που πραγματικά χρειάζονται κονδύλια. Και στη νέα περίοδο προγραμματισμού αναθεωρήσαμε τον τρόπο με τον οποίο ζητούμε ενημέρωση από τα κράτη-μέλη για τις δαπάνες. Ζητήσαμε ε, να χρησιμοποιήσουν ένα νέο εναρμονισμένο κωδικό, το βαθμό της αστιφιλίας. Και γίνεται πια με εναρμονισμένο τρόπο της αστικοποίησης μάλλον. Έτσι, με βάση το βαθμό αστικοποίησης ε, ε, διαπιστώνουμε πόσα κονδύλια αφιερώθηκαν στις πόλεις, ε, στα αστικά κέντρα, στις μικρότερες πόλεις και στην Ήπεθρο. Και το πλεονέκτημα αυτής της αλλαγής είναι ότι όχι απλώς ξέρουμε πού πηγαίνουν τα κονδύλια, αλλά πού βρίσκονται, πόσοι διαμένουν εκεί, τι ποσοστά ανεργίας, φτώχειας, παιδείας έχουν. Έτσι βλέπουμε που θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις ενισχύσεις ε, σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτά και σας ευχαριστώ γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και πολύ άρτια η έκθεση γιατί πραγματικά θίγει τα μείζωνα ζητήματα της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντόιτς, θέλετε να πάρετε και πάρετε το λόγο για μια πολύ σύντομη απάντηση. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι λακωνικός. Τόσο λακωνικός που θα είναι και σχεδόν αγένεια, διότι οι συνάδελφοι και οι προσκεκλημένοι μας ε, είπαν πάρα πολλά και πολύ σημαντικά ε, και χρήσιμα πράγματα. Δεν θα ήθελα να είμαι ευγενής απλώς και μόνο για τους τύπους. Απλώς ε, να πω ότι η σημερινή ανταλλαγή απόψεων ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και θεωρώ ότι είναι και πολλά υποσχόμενη, διότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση ε, και ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρώ να σας πω ότι δεν παραπονιέμαι, αλλά ε, φαντάζομαι ότι όλοι αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι το πρόβλημα ε, γνωμοδοτήσεων ε, όπως η δική μου είναι το γεγονός ότι είναι περιορισμένη η έκταση μιας γνωμοδότησης. Αν είχα τη δυνατότητα, θα είχα γράψει ένα έγγραφο το οποίο θα ήταν πολύ πιο μακροσκελές και έτσι θα μπορούσα ίσως να επικεντρωθώ και σε πιο σημαντικά ζητήματα. Προφανώς ε, υπάρχει δυνατότητα να προσθέσουμε κάποια σημαντικά στοιχεία σε αυτό το έγγραφο ε, μέσω τροπολογιών ε, όταν θεωρούμε ότι κάτι δεν έχει τονιστεί δεόντως ή αν θέλουμε να προσθέσουμε κάποια στοιχεία. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία πάρα πολύ ε, σύντομα σχόλια. Συμφωνώ απολύτως ε, με την Πρόεδρο και με τον κύριο Ρούι ότι δεν συζητούμε μόνο την πολιτική συνοχή και το σχέδιο Γιούνκερ εδώ, συζητούμε όλες τις πολιτικές και τη πολιτική συνοχή θα πρέπει να εναρμονιστεί θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να βρούμε συνέργειες και ίσως και πού μπορούμε να προσθέσουμε και κάποια πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρόκειται για μία προσέγγιση ε, με την οποία συμφωνούν όλοι. Δεύτερον, η ευελιξία και οι διάφορες θεματικές ενότητες. Νομίζω ότι ο κύριος Ρουίλ και η κυρία Κρέιλ Κρέλ ως συγητές ασχολήθηκαν με τα θέματα αυτά ήδη στον προηγούμενο κύκλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εστίες σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, αλλά όσον αφορά την ευελιξία... Uh, αυτό είναι πολύ σημαντικό για, κυρίως για περιοχές οι οποίες υστερούν. Ιδίως για ε, περιοχές οι οποίες βρίσκονται ε, σε πιο ε, περιφερειακές ε, ζώνες. Για την ενεργεία των νέων, σίγουρα πρόκειται για ένα φαινόμενο που πρέπει να καταπολεμήσουμε και πρέπει να βρούμε τρόπους να ε, χρησιμοποιήσουμε κονδύλια από το Ταμείο συνοχή. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στην εγγύηση για την νεολαία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, για να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο, συμφωνώ ως προς το γεγονός ότι πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, αλλά δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο σε αυτό και να αποκλείσουμε όλες τις άλλες δυνατότητες. Κατ' όλη η πολιτική συνοχής και το σχέδιο ε, Juncker θα πρέπει να εξεταστούν κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πλήρως. Σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύτιμα σχόλιά σας και αναμένω τις τροπολογίες σας και ελπίζω ότι το Μάιο θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε το κείμενο με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 5η 12 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι, για την γνωμοδότηση για την έκτη έκθεση συνοχής. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ε, το Επόμενο τμήμα της συνεδρίασής μας είναι αφιερωμένο στην ε, ε, πολιτική, ε, στην αστική πολιτική. Η συγγήτρια είναι η κυρία Κέρστιν Βέστφαλ. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων ζουν σε αστικές περιοχές και επομένως οι πόλεις αποτελούν τη ρεχοκοκονιά της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Ε, πολλές πολιτικές σε εθνικό επίπεδο έχουν ουσιαστική επιρροή στις πόλεις ή βασίζονται στα δημοτικά συμβούλια για την εφαρμογή τους επιτόπου. Οι πολιτικές ε, ε, σε διάφορους τομείς και οι ευρωπαϊκές πολιτικές πολύ συχνά δεν συντονίζονται καταλήλως και σε ένα ψήφισμα το 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε ε, με μια πιο κοινή προσέγγιση για τις πόλεις. Τον Ιούλιο πέρσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ε, μια ανακοίνωση για την αστική διάσταση των πολιτικών και η δική μας έκθεση αποτελεί απάντηση στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Το Δεκέμβριο η συγγήτρια, κυρία Βέστφαλ, ε, αναφέρθηκε στους αρχικούς της στόχους, έγινε μια πολύ σημαντική συζήτηση προκαταρκτικά επ' αυτού και σήμερα θα μας παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσής της. Προτείνω η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών να είναι η 5η 19 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο το τελικό σχέδιο έκθεσης και ε, έχουμε εδώ και τους κοιόδης εισηγητές, έχουμε εκπροσώπους από την Επιτροπή των Περιφερειών και υπάρχει και εκπρόσωπος της ΕΟΚΕ Και ε, στη συνέχεια, σε ένα ενδιαφέρον τμήμα τη ε, πρωινή μα συζήτηση, θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με την ομάδα Ευρωπαϊκή Πόλη και θα ε, έχουμε και μια παρουσίαση από κάποιον εκπρόσωπο του δικτύου των Ευρωπαϊκών Πόλεων. Θα είναι η πόλη του Μπουργκά στη Βουλγαρία. Καταλαβαίνετε, είναι βουλγαρικό το ζήτημα εδώ. Θα έχουμε εδώ λοιπόν τον εισηγητή, θα ακούσουμε τον εισηγητή, την άποψη των συναδέλφων, την άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών, την ε, άποψη της Ομάδας Ευρωπαϊκές Πόλεις και θα έχουμε και μια παρουσίαση από μια Ευρωπαϊκή Πόλη. Έχετε το λόγο κυρία Βέστφαλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πώς τυχαίνει, είμαι πάντα κρυολογημένη όταν πρέπει να παρουσιάσω κάτι. Ο συνάδελφος ο Ντόιτς έχει δίκιο όσον αφορά την έκταση ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο να αναπτύξουμε τα θέματά μας. Άκουσα πολλές φορές σήμερα πόσο σημαντικές είναι οι πόλεις και ότι στην πράξη υπάρχει μεγαλύτερη ελπίδα και όντως ελπίζω ότι δεν θα είναι μόνο εδώ για εμάς σημαντικές πόλεις αλλά και για τους εκπροσώπους των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων ώστε να συμπεριληφθούν στον πολιτικό σχεδιασμό του μέλλοντος. Όπως υπόθηκε, το 3% τέταρτα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ε, ε πληθυσμού ζουν σε πόλεις. Τα δύο του ΑΕΠ ε, παράγεται στις πόλεις. Το 70% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εφαρμόζεται σε ε, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι το 5% ε, των κονδυλίων του ΕΤΠΑ απορροφούνται σε τοπικό αστικό επίπεδο. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι κάποια... Ε, αυτοί είναι κάποιοι λόγοι που θα πρέπει να μας κάνουν ασχοληθούμε περισσότερο με την αστική διάσταση. Και γι' αυτό καλωσορίζω την ε, ανακοίνωση για μια αστική ημερήσια διάταξη, για μια αστική διάσταση Και θα πω αυτό που λέμε και στα γερμανικά, ότι η ελπίδα παθαίνει πάντα τελευταία. Σε συνομιλίες με την Επιτροπή των Περιφερειών και με την ΕΟΚΕ, με τα EuroCities και τους εκπροσώπους άλλων πόλεων, παρατήρησα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ενάγκη για μια αστική διάσταση. Και επίσης να καλωσορίσω τον Δήμαρχο της Δέλφτ, με τον οποίο είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα αυτό. Ο διάλογος αυτός συλλαμβάνει χώρο και στην Ευρωπαϊκή των Περιφερειών, τον κύριο Μπάρντ από την ΕΟΚΕ. Να τον ευχαριστήσω και αυτόν και πολλούς άλλους εκπροσώπους ε, του EuroCities για τις περιεκτικές συζητήσεις που κάναμε. Στη δικιά μου έκθεση κάνω κάποιες προτάσεις που είναι σημαντικές για την Επιτροπή των Περιφερειών που θα πρέπει να δώσουμε βάρος. Η αστική διάσταση θα πρέπει κατά την άποψή μου, και αυτό θέλω εξ αρχής να το τονίσω και να το αποσαφηνίσω, θα πρέπει να παρέχει ένα πλαίσιο για τις πόλεις, ε, μια εργαλειοθήκη θα λέγαμε, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια εργαλεία που θα τα εφαρμόσουν σε αστικό επίπεδο. Αυτό που δεν αναφέρω λεπτομερώς στην έκθεσή μου, ποιες είναι, τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις. Το δημογραφικό θέμα, η καινοτομία, η φτώχεια, η ανάγκη για στέγαση, οι κλιματικές αλλαγές, όλα αυτά θίγονται. Όμως, θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει ουσιαστικά αυτή η έκθεση να παρέχει αυτή την εργαλειοθήκη ώστε οι πόλεις να μπορούν να αντλήσουν δομικά στοιχεία από αυτή την εργαλειοθήκη ώστε να ε, τα αξιοποιήσουν σε αστικό επίπεδο. Στο πρώτο σημείο της μέσης διάταξης σήμερα άκουσαμε πολλές φορές τον όρο πόλη. δεν είναι μια πολιτική που αφορά αποκλειστικά τις μεγάλες πόλεις. Αφορά τις μικρότερες, τις μεσαίες και μεγαλύτερες πόλεις. Εγώ προέρχομαι από μια πόλη 50.000 κατοίκων, παραδείγματος χάρη. Αλλά αναφερόμαστε και στις ευρύτερες λειτουργικές αστικές περιοχές. Θέλω μια αστική πολιτική η οποία θα περιλαμβάνει και τις γύρω περιοχές, γιατί δεν μπορεί να ενωθεί το ένα χωρίς το άλλο. Η αστική διάσταση θα, πρέπει, θα αποτελεί συστατικό, απαραίτητο συστατικό για πολλές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα σε κάποια σημεία της εκθεσής μου. Ε, πρώτον, θεωρώ ότι αυτό που αναφέρουμε τα τελευταία πέντε χρόνια, οι πόλεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν με πιο κατάλληλο τρόπο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό το είδαμε και στην ε, διαμόρφωση διαφορετικών ε, ταμείων. Η αρχή της εταιρική σχέσης. Θα πρέπει εγκαίρως να συμπεριληφθούν οι πόλεις Να εφαρμοστεί δηλαδή αυτή η αρχή της εταιρικής σχέσης Υπόθηκε νωρίτερα ότι αυτό δεν το επιθυμούσαν τα κράτη-μέλη μου. αυτό, αυτό το κομμάτι είναι ζωτική σημασία, ε, το κομμάτι τη εταιρική σχέση. Αυτή η αρχή σε κάποια κράτη-μέλη είχε εφαρμοστεί, σε κάποια άλλα καθόλου. Έτσι λοιπόν όχι μόνο εμεί, αλλά και τα άλλα θεσμικά όργανα θα πρέπει να φροντίσουν αυτή η αρχή τη εταιρική σχέσης να ε, μπορεί να είναι και βιώσιμη. θα πρέπει επομένως να υπάρχει έγκυρη εμπλοκή των ε, τοπικών ε, αρχών. Αυτό που φοβίζει της πόλης είναι οι αντιφατικές ε, προδιαρθές από τις ε, Βρυξέλλες και η δυσκολία εφαρμογής. Αν αυτό το αποφύγουμε εκ των προτέρων, τότε στην πράξη θα έχουμε κερδίσει πολλά σε επίπεδο ευρωπαϊκή πολιτικής. Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι πρέπει σε κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία να συμπεριλαμβάνουμε και τις πόλεις και να τι λαμβάνουμε υπόψη κλιματική αλλαγή, επενδύσεις και τα λοιπά, καινοτομία, αυτά όλα αφορούν πάντοτε τις πόλεις. Θα πρέπει τις πόλεις να τις λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε τομέα της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν να έχουμε μια καλύτερη μέθοδο συνεργασίας ώστε να υπάρχει συνοχή ε, ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα. Προτείνω και μια μελέτη αντικτύπου, εδαφική μελέτη αντικτύπου, και όσον αφορά τα ταμεία και τα κονδύλια, θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη και σε αυτό το σημείο της πόλης. Η παροχή πολλών διαφορετικών δυνατοτήτων χρηματοδότηση, πολλή Θα πρέπει παράλληλα να έχουμε συνέργεια μεταξύ των ταμείων, ώστε οι πόλεις να μπορούν να βρουν ε, λύσεις κομμένες στα μέτρα τους. Και κατά τρίτον, και κάτι πολύ σημαντικό, όταν κάνουμε λόγο για τις πόλεις, τις λαμβάνουμε υπόψη, θα πρέπει αυτή η συμπερίληψη των πόλεων να θεσμοποιηθεί, να θεσμοθετηθεί μάλλον. Όμως αυτό είναι καθοριστικό, να τις λαμβάνουμε υπόψη. Σε αυτό το κομμάτι δεν έχουν γίνει πολλά τελευταία χρόνια και θα πρέπει στην πράξη να προωθήσουμε ίσως και μια αλλαγή του συστήματος. Να υπάρχει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών ε, τομέων της πολιτικής, ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα για τις πόλεις. Φυσικά στο Κοινοβούλιο, ε, στο Urban Group έχουμε κάνει αναφορά σε αυτό στην περίληψη των πόλεων. Όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει και το άλλο θέμα ότι στην Επιτροπή υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα. Θα πρέπει να υπάρχουν άτομα στην Επιτροπή που θα ασχολούνται αποκλειστικά με το θέμα των πόλεων. Και παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν και αποφάσεις. Αυτό το άτομο το οποίο θα είναι εντεταλμένο για θέματα πόλεων θα πρέπει να βρει ποιε είναι οι προτάσεις της Γενικής Διεύθυνσης και τι επίδραση έχουν αυτές ε, σε επίπεδο πόλεων. Το εκταλμένο άτομο αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχει και αρμοδιότητες και φυσικά και το Συμβούλιο με ε, συναντήσεις ε, με τους αρμόδιους υπουργούς για θέματα αστικά να χαράζει και σχετικές πολιτικές. Είναι ένα αφιλεγόμενο θέμα, όμως θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τις μελλοντικές εξελίξεις. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ε, για τις πόλη δεν θα πρέπει να ακολουθεί μια μέθοδο ε, top-down. Θα πρέπει να είναι και μια προσέγγιση bottom-up, από τα κάτω προς τα πάνω. Να υπάρχει μια πλατφόρμα για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των πόλεων. Με το Urbact και το δίκτυο αστικής ανάπτυξης έχει δημιουργηθεί μια πολύ καλή πλατφόρμα Υπάρχουν και θεματικά δικτύα όπως το EuroCities και το Habitat και άλλα δίκτυα δίνουν αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας. Θα πρέπει να εξελιχθούν, να αναπτυχθούν περαιτέρω αυτά τα δίκτυα και να υπάρχει καλύτερο συντονισμό μεταξύ τους. Ένα νέο μοντέλο ε, πολυπίδησης κυβέρνησης με καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών ώστε να γίνεται ανταλλαγή στατιστικών δεδομένων <coughs> ανάμεσα σε αυτά τα δίκτυα και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε από την μια πλευρά να έχουμε την κατάλληλη πληροφόρηση και από την άλλη πλευρά να χαράξουμε την ε, κατάλληλη πολιτική αγαπητοί συνάδελφοι. Κατά την άποψή μου θεωρώ ότι στην πράξη χρειαζόμαστε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για το πώς βλέπουμε και πώς θέλουμε να διαμορφώσουμε την ε, πολιτική για τις πόλεις. Περισσότερη συνοχή, σχηρότερο συντονισμός, ε, έγκαιρη συμπερίληψη των ενδιαφερόμενων ε, μερών και προσέγγιση bottom-up. Αυτά είναι τα βασικά σημεία στα οποία αναφέρομαι. Αν υπομονώ να ακούσω τις προτάσεις των συναδέλφων αλλά και των σχεδόν εισηγητών. Προσπάθησα στο σχέδιο ε, να συμπεριλάβω κάποιες προτάσεις από την τελευταία φορά, αλλά φυσικά δεν μπόρεσα ε, να τα θίξω όλα αυτά, όλες αυτές τις προτάσεις, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος Ντόιτς, έχουμε πολύ περιορισμένο, ε, είναι περιορισμένη έκταση η έκθεση, οπότε δεν μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά σε όλα. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος που έχει διεξαχθεί τον τελευταίο χρόνο για αυτό το θέμα. Να μην το αφήσουμε να φύγει από την ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Βέστφαλ. Ακούσουμε τώρα τις παρουσιάσεις των σχεδόν εισηγητών. Δεν βλέπω όμως τον κύριο Αλμπρίχτα από το ΕΛΚ, ούτε τον κύριο Λούρ, Εσά, σα είδα, σα είδα. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Βαρμίλτεμπορκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα ευρωπαϊκό αστικό θεματολόγιο. Αυτή είναι μια εξαιρετική βάση για τη συζήτηση και καλωσορίζω και τους εκπροσώπους ε, της Επιτροπής των, Περιφερειών, των Περιφερειών, τον κύριο Φερκέρκα και τους εκπροσώπους του EuroCities, της Ομάδας των Ευρωπαϊκών Πόλεων, που είναι στενοί μας συνεργάτες για να διαφαρμόσουμε ένα γνήσιο ευρωπαϊκό αστικό θεματολόγιο. Νομίζω ότι όλοι οι παρόντες είμαστε πεπισμένοι για την ανάγκη καλύτερου συντονισμού της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής για τις πόλεις θα πρέπει να διαμορφωθεί μια πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική τομεακή στις πόλεις. Βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις ε, κοινωνικές όπως αναφέρονται και στο πρόγραμμα για τον ορίζοντα του 2020 και πρέπει να προτείνουμε απτές και χειροπιαστές λύσεις. Χαίρομαι λοιπόν που συζητούμε τώρα για το Ευρωπαϊκό Αστικό Θεματολόγιο. Αυτό που μου είναι μία διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν την ανακοίνωση. Γιατί ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις. Κρίμα, γιατί θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μία σύγκληση και ένα παραλληλισμό των εργασιών μας. Γιατί εδώ και χρόνια συζητούμε το αστικό θεματολόγιο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά έχουμε μείνει στα λόγια και στη θεωρία. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, για να μην πω ότι έχουμε καθυστερήσει και όλα, για δράση. Θα ήθελα και εγώ μετά την εισηγήτρια να μιλήσω για συγκεκριμένα θέματα. Στο σημείο 20 της έκθεσης, η κυρία Βέστφαλ προτείνει να δώσουμε έμφαση σε διάφορες προτεραιότητες του αστικού θεματολογίου και ιδιαίτερα στην κοινωνική ένταξη, στη δημογραφική ανάπτυξη και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα ή αηφορία. Πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Τι γίνεται όμως με τη δημιουργία αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, γιατί πολλές πόλεις το κάνουν. Και είναι ένα θέμα που άπτεται της αηφόρου ανάπτυξης. Το 2050 θα έχουμε πολλές πόλεις που θα είναι ενεργειακά ουδέτερες, δηλαδή ε, ενεργειακά αυτάρκης. Θα παράγουν τη δική τους ενέργεια και μάλιστα με πολύ και μηδενική εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, κυρίως διοξιδίου του άνθρακα. Θεωρώ ότι οι πόλεις ε, ε, είναι θύλακες, ή κέντρα καινοτομία και ε, κινητήρια μοχλή της οικονομικής ανάπτυξης. Στα αστικά κέντρα δημιουργούνται οι υπηρεσίες που χρειαζόμαστε. Φυσικά στο θεματολόγιο θα πρέπει να κάνουμε και μία ράξη των προτεραιοτήτων μας. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Αλλά θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη. Αστική κινητικότητα. Πώς θα αποφύγουμε μια ασφυξία των πόλεων με τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις στενοπούς ε, αναζητώντας τρόπους ε, αηφόρων μεταφορών και απρόσκοπτης ε, κυκλοφορίας στο εσωτερικό των πόλεων. Συμφωνώ με την εισηγήτρια. Το θέμα της κοινωνικής ένταξης, δημογραφική ανάπτυξη, περιβαλλοντική αηφορία είναι πρωταρχική στόχη. Αλλά μας λείπει από την έκθεση μία αναφορά της πολύ ε, σημαντικής πρωτοβουλίας ε, της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης για την Καινοτομία. Smart Cities and Communities, ευφύς, πόλεις και κοινότητες. Εκεί δημιουργείται γόνιμο έδαφος ε, για τη γνώση και την καινοτομία. Και γιατί να μην εξασφαλίσουμε μία χρηματοδότηση από τον ορίζοντα 2020 για ερευνητικά προγράμματα τέτοιας φύσης. Γιατί ιδέες υπάρχουν, θα πρέπει να τις ενθαρρύνουμε και να τις χρηματοδοτήσουμε. Πρόκειται για στρα, στρατηγικές και διαρθρωτικές επενδύσεις. Επίσης, να δημιουργήσουμε πλατφόρμες γνώσης και πληροφορίας ε, για νέα σχέδια στις πόλεις. Θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλειών στην έκθεσή μας. Χρειάζεται φυσικά καλύτερο συντονισμός των ευρωπαϊκών πολιτικών. και μια αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας ακόμη και στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί που ετοιμάζονται οι προτάσεις και σχεδιάζονται τα προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η, νοοτροπία, η αλλαγή της νοοτροπίας και της κουλτούρας να ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βάζει τις βάσεις ε, της, ε, του αστικού θεματολογίου. Επίσης θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση και του εδαφικού αντικτύπου και με βάση τα πορίσματά της ίσως να αλλάξουμε και την προσέγγισή μας. Και αντί να δημιουργούμε νέες δομές, καλύτερα να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες δομές. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλό θα ήταν να στήσει μια ομάδα εργασίας που στόχο έχει να περιλαμβάνει την αστική διάσταση σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Έτσι θα εξασφαλιστεί η συνάφεια και η συνοχή. Γιατί να μην έχουμε και έναν ειδικό απεσταλμένο ή επιτετραμένο για την αστική ανάπτυξη. Έναν εμπειρογνώμονα με δεξιότητες και γνώσεις που θα ασχολείται με το θέμα αυτό. Γιατί ε, να μην αναθέσουμε αυτό το θέμα στον Επίτροπο της περιφερειακής ανάπτυξης. Να διευρύνει το φυλάκιό του και προς τις πόλεις και να συμπεριλαμβάνει την αστική διάσταση συστηματικά σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Να έχουμε έναν αρμόδιο επίτροπο ή τον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα ασχολείται και με τα θέματα της αστικής διάστασης. Επίσης, ό,τι αφορά τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. για να προλαμβάνουμε και να αποφεύγουμε τα προβλήματα. Η έγκαιρη προειδοποίηση είναι σημαντική για να μην ε, βυζαντινολογούμε με τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ουσία, το περιεχόμενο. Ενέργεια, η φόρος ανάπτυξη, οικολογία. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Και θέλουμε να βρούμε τη σωστή πορεία τη σωστή κατεύθυνση, καλό θα ήταν να προσανατολιστούμε στη βελτίωση των υπαρχουσών δομών και όχι στη δημιουργία νέων. Θέρμα παρακαλώ τους και ηγητές και τους ομιλητές που θα λάβουν το λόγο να είναι πιο λακωνικοί. Βέβαια, Ωραία, ωραία αυτή η πρόταση και το όνειρο να έχουμε έναν ειδικό συντονιστή για την αστική διάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Γιατί θεωρώ ότι η συγγήτρια έχει, μας προσφέρει μια πάρα πολύ καλή βάση. Θα έχουμε και επικοδομητικό διάλογο. Θέλω συγκεκριμένα δύο θέματα να τα κοιτάξουμε παραπάνω. Και τα οποία θα τα αναφέρω σκιώδη συγγήτρια. Κατά πρώτον, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ορίσουμε πιο με μεγαλύτερη σαφήνεια πώς θα πώς θα ορίσουμε την κατάσταση που βρίσκονται οι πόλεις. Δηλαδή, να έχουμε πιο συγκεκριμένα κριτήρια. Γιατί από την πλευρά μου... Ε, θεωρώ ότι υπάρχουν θέματα όσον αφορά την ε, πρόνοια σε τοπικό επίπεδο υπάρχει πίεση για εξοικονόμηση στο κομμάτι αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα πρέπει να μπορούμε να ε, διαπιστώσουμε και να εντοπίσουμε σε τι κατάσταση ακριβώ βρίσκονται οι πόλεις. Όσον αφορά την, ε, τον ορισμό πολιτικών στόχων, χρειάζεται μία ημερική διάταξη, ένα αστικό θεματολόγιο. Όμως το θέμα των συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να το ε, ορίσουμε πιο συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα σημεία και θα πρέπει αυτό να το λάβουμε όψη και στις ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος του κύριο Λιούερ, ο οποίος έφτασε εγκαίρος. Ευχαριστώ αυτό. Ε, είμαι σχέση σε δύο επιτροπέ την ίδια μέρα και γι' αυτό άρχισα. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια όσον αφορά ε, να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτή την ε, γνωμοδότηση. Τα ερωτήματα που υπάρχουν σε θέματα συνοχής, προβλήματα που διαρκούν δεκαετίες ολόκληρες σε κάποια κράτη-μέλη. ενώ κάποια άλλα κράτη έχουν σημειώσει βελτιώσεις. Αλλά με τις υπάρχουσες δομές θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω αυτή την έκθεση. Ε, περιλαμβάνει πολύ ε, την αρχή της επικουρικότητας, την αρχή του bottom-up ε, κατά κύριο λόγο και όχι τόσο του από πάνω προς τη βάση. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες προσεγγίσεις ε, top-down, φεντεραλιστικές, οι οποίες ε, uh, ίσως δεν είναι και τόσο ευπρόσδεκτες, αλλά ε, λαμβάνεται αρκετά υπόψη η αρχή της επικουρικότητας, Οι παράγραφοι 23, 24 και 25, δημιουργούν την ανάγκη για νέες γραφειοκρατικές δομές ουσιαστικά καταργούνται άλλες εξωτερικές δομές και ε, από αυτές ε, έτσι λοιπόν έχουμε μεγαλύτερη επικάλυψη ενδεχομένω, περισσότερη γραφειοκρατία. Όλα αυτά δεν τα χρειαζόμαστε. Ίσως αυτές οι παράγραφοι 23 με 25 θα μπορούσαν να αφορούν την αντικατάσταση κάποιων ε, ε, μεθόδων λειτουργίας και όχι την προσθήκη. Αν και στα υπόλοιπα τμήματα ε, συμφωνώ με τα περισσότερα σχόλια που έχουν γίνει. Ευχαριστώ κύριε, Πρό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Βάν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την συγγήτρια για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Δεν είναι πρώτη φορά φυσικά που μιλάμε για τη σημασία των πόλων σε αυτή την Επιτροπή, ούτε πρώτη έκθεση αυτής της Επιτροπής για αυτό το θέμα. Έχουν γίνει προεργασίες εδώ και χρόνια, είμαι νέο μέλος, αλλά με έχει εντυπωσιάσει ήδη το πόσο πολύ ασχοληθεί με αυτό το θέμα της αστικής, του αστικού θεματολογίου. Πολύ καλή βάση έκθεση για την αστική διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Μας ε, ικανοποιεί πολύ προσέγγιση της αστικής διάστασης που θα πρέπει να ε, γίνει, ε, να ενταχθεί και να οριστούν οι αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων. Συμφωνούμε με όλα αυτά. Όμω θα πω ότι μα λείπουν και εμά κάποια βασικά στοιχεία, όπω είπε και η προλαλήσασα. Θέματα που συζήτησαμε το Δεκέμβριο Είπατε ότι έχετε κάποιους περιορισμούς ως προς το περιεχόμενο και ότι δεν συμπεριλάβατε τα κριτήρια και το πλαίσιο, το γενικότερο για τις πόλεις για λόγους ε, ε, περιορισμού. Όμως πιστεύω ότι μία έκθεση που αφορά την αστική διάσταση θα πρέπει να συμπεριλάβει μια κοινή ανάλυση και έναν ορισμό όπως υποστήριξε και ο συνάδελφος των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις, ε, κλιματική αλλαγή, φτώχεια, έλλειψη στέγας κτλ. Το θέμα της ε, ανεργίας, ε, της αγοράς εργασίας, θα πρέπει και αυτό να συμπεριληφθεί. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά κατά την μου και οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες θα πρέπει επομένως αυτό το πλαίσιο να καθοριστεί πιο συγκεκριμένα γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ και με την ε, ε, πολιτική φιλελευθεροποίηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε όλα αυτά, επομένω, από μια έκθεση που αφορά ε, στο ρόλο των πόλεων σε μια κοινή Ευρώπη. Ειδικά οι τομεί που ε, θίγονται άμεσα από την ευρωπαϊκή πολιτική, αυτοί οι τομεί θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή την έκθεση. Έγινε λόγος για το Ευρώπη 2020. Όμως δεν περιλαμβάνει μόνο την ε, κλιματική αλλαγή, την ε, ισότητα των φύλων, ε, την κλιματική αλλαγή όπως είπαμε και πριν, την φτώχεια κτλ. Όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν και να συμπεριληφθούν εδώ παράλληλα με την περιορισμένη χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι χώρες και αυτό το περιορισμένο εφημισμός πρέπει να πω. Αυτή η πολιτική περικοπών γενικά που έχει επηρεάσει και αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά όταν μιλάμε για τις μελλοντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι πόλεις και από την πλευρά μας στο Κοινοβούλιο πρέπει ε, να τα συμπεριλάβουμε αυτά. Θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτή την ε, αστική διάσταση. Κάνετε λόγο ε, για τη δημοκρατική διάσταση, την προσέγγιση bottom-up. Το αναφέρετε, αλλά θέλουμε να το τονίσετε ακόμα περισσότερο. Να τονίσετε περισσότερο ρόλο στις κοινωνίας των πολιτών και το να δημιουργηθεί ένας διάλογος σε μια αστική, ε, για ένα αστικό θεματολόγιο. Οι κατευθυντήρε γραμμές που μα δόθηκαν το ευρωπαϊκό εξάμεινο για την κοινωνία των πολιτών να συμπεριληφθούν δηλαδή και εδώ στο θέμα της αστική διάσταση ε, τη ευρωπαϊκή πολιτικής, των ευρωπαϊκών πολιτικών. Και να γίνει και μια αναφορά στα διευθυντικά ταμεία στην, ε, ε, στο θέμα στην πολιτική των επενδύσεων. Θα πρέπει να γίνει και σε αυτό αναφορά και στι προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε με το ε, σχέδιο επενδύσεων. όπου περιλαμβάνονται οι πόλης, αλλά δεν υπάρχει σαφής ε, αναφορά της αρχής ε, της εταιρική σχέσης με την εμπλοκή των τοπικών και περιφερειακών ε, αρχών. Θεωρώ ότι και αυτό θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτή την έκθεση. Θα ήθελα λοιπόν λοιπόν ε, να συμπληρωθούν όλα αυτά σε ενδεχόμενε τροπολογίε. Νομίζω μέχρι τις 13 Μαρτίου είπατε ότι είναι προθεσμία. Και να γίνει αναφορά στις μετροπολιτικές περιοχές, κάτι που δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ. Όπως είπα όμως και πριν, είναι πολύ καλή η βάση που μας προσφέρει η συγγήτρια και θα πρέπει να ε, γίνει αναφορά συγκεκριμένη στις ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις και στην κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα την έκθεση τη συναδέλφου και να σταθώ σε τρία σημεία της έκθεσή τη. Πρώτον, η ανάγκη υποστήριξη των ολοκληρωμένων εδαφικών στρατηγικών μέσω κανόνων και κοινού στρατηγικού σχεδιασμού. Δεύτερον, όσον αφορά τη σημασία τη ε, ε, παρακίνηση προ τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούνται μέσα όπω το CLLD και το ET. Επίσης, ε, ε, το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει δήλωση προθέσεων, η, η συμμετοχή όμως ε, πόλεων στον προγραμματισμό για το 2014-2020 ήταν αρκετά μικρή. Να κάνω κάποιες προτάσεις τώρα. Το θέμα της ε, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, της επικουρικότητας, της αρχής της εταιρικής σχέσης ε, υπενθυμίζεται και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην έκθεση της συναδέλφου. Και θα πρέπει να επισημάνω κι εγώ ότι αυτό είναι ε, βασική αρχή της προγραμματικής περίοδου και της ίδιας της πολιτικής συνοχής. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να τονίσουμε στα πλαίσια μιας πραγματικής συμμετοχής στο αστικό πλαίσιο τη σημασία μιας συμμετοχής όλων των τοπικών φορέων και όχι μόνο τους εκπροσώπους ε, των Δήμων, αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό κατά την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Σε κάποιες περιοχές δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ε, υπήρξε και σχετική ερώτηση επί του ζητήματος και παρά τις διαβεβαιώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων, ε, των οικονομικών, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων θα γινόταν όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, είχαμε αρκετές υποδείξεις επιτόπου από διάφορες περιοχές ότι ε, στην πραγματικότητα αναφέρονται απλώς σε μια τυπική συμμετοχή χωρίς καμία προστιθέμενη αξία. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να προτείνω ε, σχετίζεται και με την ε, έκθεση για τις ευρωπαϊκές πόλεις για το 2014 και σχετίζεται με το γεγονός ότι μία αστική πολιτική δεν μπορεί να αφορά αποκλειστικά και μόνο πόλεις. Μόνο μια εναρμονική σχέση μεταξύ πόλεων και των γύρω περιοχών, κυρίως όταν πρόκειται για, της, ε, για περιοχές της μπορεί να βοηθήσει να έχουμε πραγματική συνεισφορά στην εδαφική συνιστόσα και στην περιφερειακή συνέχεια. Ολοκληρώνοντας να παρατηρήσω ότι στην έκθεση της συναδέλφου δεν ε, βλέπω κάποια συγκεκριμένη μνήμα σε ένα πρόβλημα κατά την άποψή μου ουσιαστικό. Το θέμα της ε, ε, αστικής αναγέννησης, ένα θέμα το οποίο είχα υποβάλει και στην ανταλλαγή απόψεων που κάναμε στην συζήτηση του Δεκεμβρίου και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διάφορα σημεία στην έκθεση της συζυγήτριας αναφέρουν τις πόλους ως κινητήριο μοχλό αλλαγών και ολοκλήρωσης και σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Επομένως, ε, και επειδή ακριβώ ε, προβλέπεται ότι θα υπάρξει δημογραφική αύξηση στις πόλεις από τώρα μέχρι το 2060, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές για να αναβιώσουμε τα ιστορικά κέντρα πολλών πόλεων και να ε, δίνουμε αντικίνητρα για την κατασκευή κτηρίων σε κάποιες περιοχές οι οποίες πολύ συχνά δεν έχουν και καλή σύνδεση με το κέντρο της πόλης και μετατρέπονται σε γκέτο. Ε, και επειδή αναφερόμαστε και στον εγκάσιο χαρακτήρα των κοινωνικών και πολιτιστικών ε, πτυχών, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στο πλαίσιο των πόλεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε με τις ε, απόψεις των σχεδόν εισηγητών και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζέλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την συνάδελφο Βέσφαλ για την περιεκτική έκθεση για την αστική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βρισκόμαστε σε ένα κέριο σημείο πριν από πέντε χρόνια όταν μπήκα στο κοινοβούλιο Άκουσα από πολλούς συναδέλφους ότι οι πόλεις είναι κομμάτι της επικουρικότητα, ότι δεν έχουν ε, πολύ μεγάλη σχέση με την Ευρώπη και το πιο σημαντικά θέμα είναι η γεωργία, η αλληλεία κτλ. Και αυτό, αυτή η προσέγγιση συνεχίστηκε Αναφέρθηκε πριν από τους συναδέλφους ότι βασικός τόπος κατοικίας των ε, πολιτών της Ευρώπης είναι η πόλη. Και δεν υπάρχει ένεδος πόλης. Έχουμε τις μικρές, μεσαίες, μεγάλες πόλεις. Στο Βερολίνο έχουν εισέλθει πλέον 40 με 50.000 ε, νέοι κάτοικοι. Αυτό όμως φυσικά δημιουργεί προβλήματα σε θέματα υποδομών, παροχή στέγασης κτλ. Έχουμε κάποιες μεσαίες μικρές πόλεις οι οποίες ε, έχουν δημογραφικά προβλήματα γιατί πολλοί φεύγουν από εκεί και όλα αυτά φυσικά σχετίζονται με, την, ε, με τους στόχους ε, της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και φυσικά έχει περάσει το μισό διάστημα, το μισό χρονικό διάστημα, οπότε πρέπει να δούμε σε ποιο επίπεδο έχουμε φτάσει ως προς την επιτεύξη αυτών των στόχων. Όταν η στοχοθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο, εκεί που ζουν οι πολίτες της Ευρώπης, τότε δεν θα μπορέσουν φυσικά να οδηγήσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την έκθεση. Αυτό που πετύχαμε τα πέντε τελευταία χρόνια σε αυτή την Επιτροπή είναι η αστική διάσταση να αποτελέσει κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτικής και να μείνει στις συνειδήσεις μας, να γίνουμε συνειδητοί ως προς αυτό. Όσον αφορά την εταιρική σχέση και τα επιχειρησικά προγράμματα, πιστεύω ότι σε αυτά τα δύο τα θέματα υπολείπεται η πολιτική για τις πόλεις. Γίνεται χρήση των διευθυντικών ταμείων για την ε, επίτευξη ε, προσωπικών στόχων, όμως σε άλλα σε σχέση με άλλους ε, τομείς ε, ε, δεν λαμβάνεται και τόσο πολύ υπόψη η πόλη. Με αυτή την έκθεση έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε συνειδητοί ως προς την ανάγκη συμπερίληψης του, ε, του διάταξης ε, στην ευρωπαϊκή πολιτική και να δημιουργήσουμε σύνδεσμο, ε, να συνδυάσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική με την τοπική διάσταση. ώστε η συμβίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει ε, κέντρο βάρους στις συζητήσεις, στις συζητήσεις μας. και ότι όταν κάτι δεν ε, βιώνεται πρώτα στο τοπικό επίπεδο, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εφαρμόσουμε αυτό το ε, ευρωπαϊκό ειδόδες που φανταζόμαστε. είναι θέματα που τα συζητάμε και σε άλλες επιτροπές σε σχέση με την απασχόληση, τη μετανάστευση, την ανάπτυξη. Πρέπει να δούμε πού παρουσιάζονται τα προβλήματα. Και να δούμε σε ποιους τομείς πρέπει να χαράξουμε πολιτική, πολιτικές. υπάρχει στήριξη από πλευρά μα και γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε και αυτή την έκθεση και τι πτυχέ τι οποίε αναφέρεται. Και σίγουρα η κυρία Βέσφαλ μας δίνει μια πολύ καλή βάση, γιατί το θέμα α, το θέμα των πόλων θα πρέπει να συζητηθεί στην Ολομέλεια αλλά σε μια κέρια στιγμή που θα τραβήξει και την προσοχή όλων και της ε, δημοσιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα τελευταίος ομιλητής ο κύριος Φανίστερ Ρόι. Σας ευχαριστώ. Επανέρχομαι στο τελευταίο σχόλιο. Για την πρόταση αυτή θα πρέπει να γίνει εκτενή συζήτηση στην Ολομέλεια επ' ευκαιρία και της έκτης έκθεσης συνοχής. Γιατί είναι κρίμα να υποβάλλουμε συζητήσεις χωρίς να αναπτύσσονται σε μια συζήτηση. Κάτι τέτοιο απαξιώνει το έργο μας. Επίσης, Θέλουμε συζήτηση για τη συνοχή, γιατί όταν μιλάμε για συνοχή, εννοείται ότι μιλάμε και για τις πόλεις. Από την έκθεση λείπουν κάποιοι εδαφικοί στόχοι. Γιατί αν θέλουμε να προωθήσουμε την αστική διάσταση και τις πόλεις και να τις φέρουμε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης, θα πρέπει να εγγύψουμε και στους εδαφικούς στόχους. Βέβαια οι πόλεις ε, είναι αναπόσπαστο τμήμα των χωρών μελών, ανήκουν στη γεωγραφική τους επικράτεια και εντάσσονται φυσικά και στις περιφέρειες. Και βλέπουμε τις, την κατάσταση, την οικονομική, κοινωνική κατάσταση και τις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών. Ανισότητες υπάρχουν όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό και μιλούμε για πολύ επίπεδη διακυβέρνηση. Και οι ευρωπαϊκές συνθήκες ε, προβλέπουν δράσεις όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ας μην ξεχνούμε αυτές τις σημαντικές ε, διαστάσεις που δυστυχώς ε, δεν αναπτύσσονται δεόντως ή δεν αξιοποιούνται δεόντως. Και φυσικά, μια και μιλάμε για συνοχή και έκθεση συνοχής, δεν μπορούμε παρά να παραπέμπουμε το θέμα και στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαπιστώνουμε ότι η θεωρία είναι καλή, τα λόγια είναι ευάρεστα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει συνέχεια στα έργα. Η, προεδρία, η προηγούμενη Προεδρία έχει υποβάλει στο Συμβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, επαναφορά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης του αστικού θεματολογίου. Είναι σημαντική αυτή η προσοχή που είχε δώσει το τελευταίο Συμβούλιο στο θέμα αυτό. Πώς λοιπόν θα προχωρήσουμε. Ζητήσαμε έναν ειδικό συντονιστή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αστική διάσταση. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή μεθοδολογία. Και δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο, γιατί είναι λεπτό το ζήτημα. Έχουμε το θεσμό των EuroCities, ε, της ομάδας των Ευρωπαϊκών Πόλεων, εδώ και 20 χρόνια. Οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι πολύ καλοί συνομιλητές μας και θα πρέπει να ακούμε τη φωνή τους. Επίσης, καλό θα ήταν να έχουν και οι ευρωπαϊκές πόλεις άμεσες απευθείας επαφές με, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει ένας απολογισμός της κατάστασης και να βελτιωθεί και το modus operandi, η μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί να μην συνάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εταιρική σχέση με τις ευρωπαϊκές πόλεις. Θα πρέπει να το ζητήσουν και οι ίδιες οι ευρωπαϊκές πόλεις και να παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνάψει τέτοιες εταιρικέ σχέσεις μαζί τους. Γιατί σε τελική ανάλυση οι πόλεις εφαρμόζουν ε, σε τοπικό επίπεδο την ευρωπαϊκή πολιτική. Στο παρελθόν είχαμε μεγάλες καθυστερήσεις. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να ανασκομποθούμε. Και γιατί όχι να μην ε, συνάψουμε ένα νέο σύμβολο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να οριστεί ένας νέος επιτετραμένος εκπρόσωπος συντονιστής, όπως θέλετε πείτε τον, αλλά κάποιος αρμόδιος για να επαναφέρει το αστικό θεματολόγιο και την αστική διάσταση στο επίκεντρο της συζήτησης. Θέλουμε να γίνει προτεραιότητα, όπως είχε αναγγείλει και η Ολλανδική Προεδρία στο δικό της πρόγραμμα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πολλά επίπεδα. Αλλά γιατί να μην έχουμε διασύνδεση των διαφόρων επίπεδων και το κατώτερο επίπεδο που είναι η πόλη να έχει άμεση συζήτηση με το ανώτερο επίπεδο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Πρόεδρος, αν θέλετε να δώσουμε χρόνο και να ακούσουμε και τις ευρωπαϊκές πόλεις, θα πρέπει να είστε λίγο πιο λακωνικοί στις δικές σας παρεμβάσεις. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φερκέρκ, που εκπροσωπεί την Επιτροπή των Περιφερειών και εισηγητής της γνωμοδότησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ίδιο θέμα. Είναι μάλιστα και δήμαρχος της πόλης του Ντέλφ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, οι φίλοι των πόλεων και της Ευρώπης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ σήμερα ε, στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης ως ε, εισηγητής της Επιτροπής των Περιφερειών ε, για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για ε, κυρίως το θέμα αυτό, την αστική διάσταση και τις ευρωπαϊκές πολιτικές, η Επιτροπή των Περιφερειών είναι πολύ ικανοποιημένη με τη σημασία που προσδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό. Οι πόλεις και οι αστικές περιοχές είναι μεγάλη σημασία για την Ευρώπη και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και να προσπαθήσουμε να το εντάξουμε λίγο καλύτερα στην ευρωπαϊκή χάραξη πολιτικής και ε, στην ευρωπαϊκή ε, εκπόνηση νομοθεσίας. Να συγχαρώ την εισηγήτρια για το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης, ε, την κυρία Βέσταλ. Ε, διαπιστώνει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των πόλεων στις ευρωπαϊκές πολιτικές και χαίρομαι διότι μπορώ να την προσμετρώ σύμμαχό μας για να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε εξορθολογισμό στις αστικές ε, ε, πολιτικές και στη νομοθεσία. Εγώ είμαι δήμαρχος μιας μικρής πόλης μεσαίου μεγέθους, 100.000 κατοίκων, και είμαι τμήμα της Μητροπολιτικής Περιοχής της Χάγης που έχει περίπου 3 εκατομμύρια κατοίκους. Γνωρίζω λοιπόν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να υπάρχει μια πόλη μεσαίου μεγέθους η οποία περιβάλλεται από δύο μεγαλύτερες πόλεις και υπάρχουν και μικρότερες κομμοπόλεις. Είναι λοιπόν ε, αυτό το οποίο διαπιστώνεται όχι μόνο στην, ε, ε, στις κατοχώρες αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε μικρότερες πόλεις, μεγαλύτερες πόλεις ε, πολύ μεγάλες πόλεις και όλες αυτές ε, διαδρούν μεταξύ τους και μοιράζονται και δανείζονται ε, πολιτικές και μεγέθη. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στις πόλεις. Χρειαζόμαστε ένα αστικό θεματολόγιο. Απολύτως. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δεν υπάρχει αστικό θεματολόγιο μέχρι τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία. Η Ευρώπη χρειάζεται τις πόλεις της σήμερα σε μια ε, οικονομία η οποία ε, ε, κυρίως ε, στοχεύει προς ανάπτυξη ε, και οι πόλεις είναι αυτές οι οποίες θα μας βοηθήσουμε. Ναι, στην πόλη έχουμε καινοτομία, στις πόλεις έχουμε κοινωνική συνοχή, σε αυτές τις πόλεις και στις αστικές περιοχές. Ε, ένα αστικό θεματολόγιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα αναγνωρίσει τη σημασία των πόλεων ε, και για την επίτευξη ε, των ευρωπαϊκών πολιτικών και για να μπορέσουμε να είμαστε και πιο ανταγωνιστικοί σε ευρύτερο επίπεδο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε ολοκλήρωση της αστικής διάστασης στην ευρωπαϊκή χάραξη πολιτικής και η χάραξη πολιτικής μεταφράζεται σε κανονισμούς και κανόνες και δεν αφορά μόνο την εδαφική συνοχή και τη χρηματοδότηση, αλλά ε, σημαίνει επίσης εκπόνηση νομοθεσίας, εφαρμογή νομοθεσίας και νομοθεσία με έναν τρόπο που οι πόλεις να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Αυτό εννοούσε και η κυρία Βέσφαλ με ένα σύστημα εγκυρές προειδοποίησης. Ορισμένες φορές οι πόλεις στην Ευρώπη ε, περνούν απαρατήρητε στο ανώτερο ευρωπαϊκό επίπεδο και επομένω οι πόλοι και οι εκπρόσωποι τους μπορούν να το φέρουν αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ενημερώσουν εγκαίρως ότι αυτή είναι μια νέα τάση, είναι μια νέα ε, εξέλιξη και ίσως ε, ε, αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή πολιτική στην πράξη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το σύστημα εγκαιρής προειδοποίησης. Και θα ήθελα να σταθώ και σε δύο πρόσφατες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή πολιτική. Καταρχάς, η λειτουργική όλη και τα, οι συλλογικές ομαδικές δράσεις και επίσης η τοπική κοινωνία και πολιτική. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένε δομές οι οποίες θα είναι δημιουργημένες ε, γύρω από μικρές, ε, μεσαίου μεγέθου και μεγάλε πόλεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι γνωρίζω δήμους που έχουν 100.000 κατοίκους, αλλά δεν ε, δρούν ω πόλη. Είναι απλώς μια συστάδα σπιτιών χωρίς να θεωρούνται πόλη και γνωρίζω πόλεις στην Ευρώπη 10.000 κατοίκων που πραγματικά ε, ε, συμπεριφέρονται ως πόλεις ε, και για τους πολίτες τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις ευρύτερες περιοχές τους. Θεωρώ λοιπόν ότι το μέγεθος δεν τα λέει όλα. Δεν μπορώ να πω ότι το μέγεθος δεν έχει σημασία, αλλά υπάρχουν διαφορετικές πόλεις Ε, και υπάρχουν περιοχές οι οποίες συμπεριφέρονται ως πόλεις χωρίς να λάβουμε υπόψη τον αριθμό των κατοίκων τους. Και επομένως θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο όλων αυτών των πόλεων και να, το, και να τις βοηθήσουμε. Οι πόλεις και οι κομοπόλεις συνεργάζονται με άλλες πόλεις και με την Ήπεθρο. Η Ήπεθρος είναι πάρα πολύ σημαντική για τις πόλεις για να μπορέσουν και αυτές να διαδραματίσουν σωστά το ρόλο τους. Εντός λοιπόν αυτής της συνεργασίας... Ε, οι γειτονικέ περιοχές ε, έχουν μεγάλες δυνατότητες καινοτομίας και υπάρχουν ε, φοβερές δυνατότητες και επίσης ε, αυτές οι λειτουργικές περιοχές χρειάζονται μια διαφορετική διακυβέρνηση και ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης. Οι πόλεις, όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011, αναγνωρίζεται ότι θα πρέπει να έχουν πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις περιοχές αυτές σε επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών. Αυτό όμως ακόμα δεν έχει συμπεριληφθεί στη χάραξη πολιτικής. Μια δεύτερη παρατήρηση. Διαπιστώνουμε ότι αλλάζει η σχέση μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνίας και αυτό το νιώθουμε ε, και το νιώθουμε ως πολίτες ε, στο πιο χαμηλό επίπεδο, μέσω της ε, ψηφιοποίησης της κοινωνίας, ε, της πληροφορίας και επικοινωνίας του διαδικτύου. Οι πόλεις έχουν περισσότερες απαιτήσει, αλλά έχουν και περισσότερο ισχύ. Και βλέπουμε ότι οι επιχειρηματίες ανησυχούν όλο ένα και περισσότερο για την κοινωνική τους ευθύνη. Και τέλος, οι πόλεις και οι κομοπόλεις συνεργάζονται στενά με ένα τετραπλό έλικα, δηλαδή το συνδυασμό τεσσάρων ομάδων. Έχουμε επιχειρήσεις και αγορές, ε, επιστήμη και παιδεία, κυβέρνηση και ένα τέταρτο στοιχείο που είναι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Όλο ένα και περισσότερο λοιπόν αυτέ οι τέσσερι ομάδε συνεργάζονται και δημιουργούν μια πόλη στην πράξη. Πρόκειται για ένα συνδυασμό, ο οποίος όμως έχει όλο ένα και πιο μικρό προϋπολογισμό σε τοπικό επίπεδο και βλέπουμε ότι η διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο υποχωρεί σε κάποιους τομείς πολιτικής. Δεν έχουμε πλέον τοπική διακυβέρνηση και αυτό φυσικά υποσκάπτει πρωτοβουλίες από τις πόλεις, τους πολίτες και τις κοινωνίες των πόλεων. Οι ε, άνθρωποι αναλαμβάνουν ε, πρωτοβουλίες μόνοι τους και τους ε, παροτρύνουμε να το κάνουμε, διότι υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις και κομμεπόλεις δρούν όλο ένα και περισσότερο ως συντονιστές και ως πλατφόρμες για τοπικές πρωτοβουλίες, ε, οι οποίες είναι ε, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των πολιτών τους. Και υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορετικές προσεγγίσεις ανά την Ευρώπη και η ιδέα ενός ενιαίου μοντέλου για να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές προκλήσεις σε τοπικό επίπεδο αρχίζει και χάνει έδαφος, δεν έχει αποτέλεσμα γιατί κάθε πόλη είναι διαφορετική και έχει διαφορετικές λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις νέες σχέσεις σε τοπικό επίπεδο και την διαφοροποίηση της προσέγγισης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Προκειμένου λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι δύο αυτές εξελίξεις θα ενταχθούν στη χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Επιτροπή των Περιφερειών καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια λευκή βίβλο. Μια λευκή βίβλο για, μια, ε, για ένα αστικό θεματολόγιο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πραγματική ένταξη και της αστικής διάστασης. Μετά από σχεδόν ε, δύο χρόνια συζητήσεων και αρκετών δηλώσεων και ε, συζητήσεων ήγηκε και η ώρα να δράσουμε. Η λευκή βίβλος αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξή στοιχεία. Καταρχάς, μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη πράξη πολιτικής θα πρέπει να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι πόλεις να μπορούν να επιτύχουν να έχουν ζωντανές και ελκυστικές πόλεις στις ευρύτερες περιοχές τους. Σας είπα προηγουμένω ότι οι περισσότερες πολιτικές και κανονισμοί εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο. Το αστικό θεματολόγιο λοιπόν δεν αφορά μόνο την εδαφική συνοχή και τη χρηματοδότηση, αλλά πολύ συγκεκριμένα την καλύτερη νομοθεσία, ορισμένες φορές λιγότερη νομοθεσία, τουλάχιστον ε, ολοκληρωμένη νομοθεσία ώστε να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε και να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για ανάπτυξη και θέση εργασία. Δεύτερον, ζητούμε μια πιο ει βάθο αστική διάσταση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή των Περιφερειών συγγνώμη, είναι ικανοποιημένοι με την ένταξη της αστικής διάκτασης στην παρούσα προγραμματική περίοδο στην πολιτική συνοχή και θα πρέπει να διασφαλίσουμε όμως ότι και στην πράξη η αστική διάσταση δεν θα λάβει λιγότερη ε, προσοχή από όσοι προτείνεται στο πρόγραμμα. Ε, οι πόλεις μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξης και αυτό γίνεται στις πόλεις, γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διευκολύνει ε, τις πόλεις και να τους δώσει τα χρηματικά μέσα για το επιτύχουν αυτό. Θα πρέπει να αποτελέσουμε πλατφόρμα για την ανταλλαγή των πρακτικών. Πολλέ πόλει συνεργάζονται με τοπικού εταίρου, με λύσει στα μέτρα του για την επίλυση των προβλημάτων και των προκλήσεών του και ορισμένε φορέ οι λύσει αυτέ γίνονται μεν στα μέτρα του, αλλά θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμε και για άλλε πόλει. Επομένω, θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσει πλατφόρμε για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, όπω για παράδειγμα τη Ήβητα, ε, αλλά και άλλε άλλες πλατφόρμες που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ακριβώς για αυτό το σκοπό. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρχει μια αποτελεσματική και πιο ολοκληρωμένη μέθοδος για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Όλα αυτά τα στοιχεία βέβαια σημαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια νέα προσέγγιση, μια νέα διακυβέρνηση σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και επομένως πρέπει να υπάρξει ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Υπάρχουν και πολιτιστικά και διαρθρωτικά στοιχεία τα οποία είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να μαθαίνουμε ένας από τον άλλον και να συνεργαζόμαστε ε, σε αυτή την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να επιμένουμε σε αυτή την προσέγγιση, διότι, και εδώ σας παραθέτω τα όσα έλεγε ο πρώην Επίτροπος για την ε, Περιφερειακή Πολιτική, ο Γιωχάνες Χάν, ο οποίος είναι ακόμα Επίτροπος, ε, ο Γιωχάνες Χάν έλεγε ότι το, το μέλλον της Ευρώπης θα σας διασχίσει στις πόλεις και αν δεν τα καταφέρουμε στις πόλεις δεν θα τα καταφέρουμε καθόλου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, εσάς και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι εδώ, αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και έχουμε ήδη καθυστερήσει, θα ήθελα να σας ζητήσω αν έχετε σχόλια να τα δώσετε στη γραμματεία γραπτός και εμείς ε, από εκεί και πέρα ε, θα τα διαβιβάσουμε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Κυρία Βέστφαλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ακούσω και την Επιτροπή. Ίσως θα πρέπει να δίνουμε περισσότερο χρόνο στην ημερησία διάταξη γιατί είχαμε δύο πολύ σημαντικά θέματα σήμερα το πρωί και θα πρέπει και το EuroCities να έχει χρόνο για να μιλήσει για το θέμα. Θεωρώ ότι η εισηγήση των σχεδόν και οι προτάσεις και τροπολογίες θα είναι πολύ ε, περιεκτικές. Μετά την υποβολή τροπολογιών υπάρχει συνάντηση με του σχεδόν εισηγητές. Όμως ήδη η συζήτηση που έγινε τώρα μπορεί να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα. Όσον αφορά τον ενταλμένο για τις πόλεις, θέλω να πω κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι υπήρξε μια μικρή παρεξήγηση σε αυτό το θέμα. Δεν σημαίνει για μια επιπρόσθετη, ένα επιπρόσθετο θεσμό. Κάνατε αναφορά στα λόγια ε, του Επιτρόπου Χάν που υποστηρίζει πολύ την πολιτική για τις πόλεις. Και θα πρέπει σε κάθε επιτροπή να δίνονται εξηγήσει για το τι σημαίνει η εφαρμογή κάθε πολιτικής ε, για, το, ε, για τις πόλεις. Άρα χρειαζόμαστε μια θέση που να έχει αρμοδιότητες κάποιον ενταλμένο, ο οποίος θα κουνεί χάρη τον κόδωνα του κινδύνου που θα λέει προσοχή ότι αυτό αφορά τις πόλεις. Και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να οριστεί μια τέτοια θέση ενός εντεταλμένου για θέματα πόλεων. Ναι, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε χρόνο και ότι χρειαζόμαστε και χρόνο στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, για να αναφερθούμε στην ε, ουσιαστικό θεματολόγιο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε ένα τέταρτο στη διάθεσή μας για να ακούσουμε τις ευρωπαϊκές πόλεις. Έχουμε εκπρόσωπο μιας πόλης που είναι ε, τμήμα του δικτύου Ευρωπαϊκές Πόλεις και θα ήθελα να ζητήσω ε, πέντε λεπτά επιπλέον από τους διερμηνείς για να έχουμε και τη δυνατότητα να ακούσουμε τα μηνύματα των Ευρωπαϊκών Πόλεων και ε, πιο συγκεκριμένα μίας εκ των πόλεων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε και δίνετε στις Ευρωπαϊκές Πόλεις να συμβάλλουν στη συζήτηση αυτή για το Ευρωπαϊκό στικό Θεματολόγιο. Ε, πάνω από 130 πόλεις συμμετέχουν στο EuroCities, οι περισσότερες πρωτεύουσες, ε, μέσω του δικτύου ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών για ευρύ φάσμα πολιτικών. Είμαστε η πολιτική πλατφόρμα και το φερέφωνο των πόλων στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό λοιπόν να διατρανώσουμε τη δέσμευση όλων των πόλεων ε, υπέρ του Ευρωπαϊκού Αστικού Θεματολογίου. Ως Γεροσύτης χαιρετίζουμε το γεγονό ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρατημέλη μας δίνουν τακτικά ευκαιρίε να συμβάλλουμε στη συζήτηση ε, τουλάχιστον αυτό συνέβη στο παρελθόν. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερω ε, που έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε και στη σημερινή σα συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Βέστφαλ για το σχέδιο εκθεσή τη, με θέμα την αστική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η έκθεση επισημαίνει τους λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό αστικό θεματολόγιο. Θα σταθώ στους τρεις από τους βασικότερους λόγους πριν περάσω στις ειδικέ μας προτάσεις. Γιατί χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό αστικό θεματολόγιο. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, γονιμοποιείται ουσιαστικά στο, στις πόλεις της. Οι ε, σωστές λειτουργικές πόλεις και μετροπολιτικές περιοχές έχουν ε, θεμελιώδη σημασία όχι για τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αλλά και για την Ευρώπη στο σύνολό τη. Επίσης έχουν ε, κέριο ρόλο και στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Ε, οι περισσότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχουν ε, αστική διάσταση σε πολλά θέματα, δημοκρατικές αλλαγές, δημογραφική πρόκληση, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές και το καθεξής. Θα πρέπει να αναγνωριστεί και η ικανότητα των ευρωπαϊκών πόλεων να υλοποιήσουν αυτές τις προτεραιότητες και να συμβάλλουν σε μια νέα όθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουμε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλειών που έχουν έμεσες ή άμεσες συνέπειες στις πόλεις. Για παράδειγμα, ε, το θέμα της απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής, ε, πολιτισμού, περιβάλλοντος, ενέργειας, ε, μεταφορών οικονομικού περιβάλλοντος. Τέτοιες πρωτοβουλίες δυστυχώ όμως δεν τη χάνουν επαρκού συντονισμού και μερικές φορές υπονομεύονται από τομεακές πολιτικές. Θέλουμε σαφέστερους και συνεπέστερους, συνεκτικότερους στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών που έχουν συνέπειες και αντίκτυπο της πόλης. Ως προς τους στόχους μας, δεν θα στηρίξουμε ένα αστικό θεματολόγιο που θα ε, αυξήσει το νομοθετικό φόρτο των πόλεων. Ήδη, όπως σας είπαμε, 70% της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, εφαρμόζεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και άρα και στις πόλεις. Θέλουμε προστιθέμενη αξία, να δώσουμε δυνατότητα στις πόλεις ε, να υλοποιήσουν τους στόχους του 2020 για βιώσιμη, έξυπνη και Ευρώπη που δεν θα αποκλεί και επίσης να συμβάλλουν στη χάραξη των πολιτικών, επίσης όρις με τα κράτη-μέλη ε, για να υιοθετούνται κατάλληλες πολιτικές. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώ εφαρμόζονται εμπράκτο όλα αυτά. Θέλουμε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Για παράδειγμα, είμαστε υπέρ της της πρότασης της έκθεσης να οριστεί ένας επιτετραμένος ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδιος για την αστική διάσταση. Έτσι θα εξασφαλιστεί συντονισμό στην πράξη και των πολιτικών και λήψη υπόψη της αστικής διάστασης. Έτσι θα πραγματοθεί και ο στόχος του εφνομοθετήν και θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει καλύτερο συντονισμό. Επίσης, ε, θέλουμε πιο συστηματική και άμεση ανάμειξη των πόλων στη χάραξη πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα καλό παράδειγμα θα ήταν η άμεση συμμετοχή των πόλων στις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Θα πρέπει να περάσουμε από στοιχειώδη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους σε πραγματική εταιρική σχέση με τις πόλεις ε, στηρίζουμε την έκκληση ε, της εισηγήτριας για τακτικές συνόδους κορυφής ε, με συμμετόχους από τις πόλεις και όλα τα επίπεδα της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής αυτοδιοίκησης. Έτσι θα συμβάλλουμε στις πολιτικές και σε τεχνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Μόνο με πραγμάτως αυτής της πολυεπίπεδης ε, διακυβέρνησης ε, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το αστικό θεματολόγιο. Και θα πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε να εμπλέξουμε τις πόλεις μας και τις κυβερνήσεις μας. Σίγουρα ένα αστικό θεματολόγιο θα πρέπει να είναι μια νέα ακόμη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σωστά η συγκεκριτή επισημαίνει ότι η Ευρώπη 2020 ήδη θέτει το πλαίσιο του αστικού θεματολογίου και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας αναπτύσσοντας ε, τους ε, υφιστάμενους μηχανισμούς. Έχουμε εντοπίσει πέντε τομείς με μεγάλες ε, ευκαιρίες και προοπτικές για τις πόλεις σε συνάφεια με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προτεραιότητες είναι οι εξής. Οι πόλεις είναι κινητήριος μοχλός θέσεων απασχόλησης και η φόρο ανάπτυξης. Πράσινες έξυπνες πόλεις ε, με αστική αναζωογόνηση, ανάπλαση και αποτελεσματικές πόλεις. Μόνο έτσι θα εφαρμόσουμε το αστικό θεματολόγιο και θα, θα το συνδυάσουμε με τις ευρωπαϊκές προκλήσεις. Θα συνδυάσουμε καλύτερα τις ε, τομεακές πολιτικές και τα πολλαπλά επίπεδα της διακυβέρνησης και θα επικεντρώσουμε την κοινοτική χρηματοδότηση εκεί που επιφέρει προστιθέμενη αξία. Μάλιστα σήμερα θα προβούμε σε μια διακήρυξη στο EuroCities για την απασχόληση, ζητώντας εταιρικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, και σε όλους τους τομείς προκειμένου να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα κοινοτικά κονδύλια και να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα της ανεργίας βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα, ε, αιτήσει και κλήσει προς την Επιτροπή σας. Για να υλοποιήσουμε το αστικό θεματολόγιο χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Ευρωβουλευτών που είναι οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά θα πρέπει να προσετεριστείτε και τους ενδιαφερομένους ε, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε από κοινού το αστικό θεματολόγιο και να συνεργαστούμε με πανεπιστημιακούς, ε, ερευνητές και επιχειρηματίες. Μαζί με τους δημάρχους ε, θα πρέπει να συνενώσουμε διάφορους τομείς και επίπεδα διακυβέρνησης, να στηρίξουμε την έρευνα για την ανέβρεση πρακτικών λύσεων στις αστικές και εδαφικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να εξυπηρετήσουμε όλους τους συμπολίτες. Εσείς ε, ε, θα καλέσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λογοδοτήσει σε περίπτωση που δεν συντονίσει καλά τις πολιτικές. Επίσης θα πρέπει να μεριμνήσετε ώστε να αποφευθεί επικάλυψη των πολιτικών. Φυσικά όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση θα πρέπει να κάνουν περισσότερα με λιγότερα κονδύλια εξαιτία τη συρρήκνωση των κρατικών δαπανών. Και πιστεύω ότι με το αστικό θεματολόγιο και την αστική διάσταση θα αξιοποιήσουμε καλύτερα όλε αυτέ τι προσπάθειε. Επίση, ε, είστε επιφορτισμένοι με την ε, έλεγχο εφαρμογή του νέου Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Και με την εταιρική σχέση και τον κώδικα συμπεριφορά. Ε, μπορούμε να δώσουμε το καλό παράδειγμα και σε άλλους τομείς πολιτικών που θα πρέπει να λάβουν υπόψη την αστική διάσταση και το αστικό θεματολόγιο. Εν κατακλείδη θα ήθελα να τονίσω ότι το αστικό θεματολόγιο δεν αφορά μόνο τις πόλεις. Οι πόλεις αντιμετωπίζουν στρατηγικές προκλήσεις ό,τι αφορά την αποσχόληση το περιβάλλον, την ανάπτυξη που ξεπερνούν τα διοικητικά και δημοτικά συμβούλια. Οι πόλεις και τα περίχωρά τους ε, είναι ε, αλληλοεξαρτημένες και θα πρέπει να συνεργαστούν για να βρουν καλύτερα τις πόλεις, ε, γιατί σωστά λειτουργούσε πόλεις θα ευνοήσουν και τα περίχωρά τους, θα είναι κινητήριος μοχλός της καινοτομίας και θα συμβάλλουν στην υλοποίηση της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνική συνοχής. Γι' αυτό και το αστικό θεματολόγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζεται μόνο στις πόλεις, αλλά αφορά την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υλοποιήσει στρατηγικούς στόχους για μια e e, ευφυή, αηφόρο Ευρώπη και κυρίως Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για την προσοχή σας και δίνω το λόγο στον συνάδελφο, τον Δήμαρχο Μπουργκάς. Ευχαριστώ την κυρία Καρίν Ντανιέλ, την ε, αντιδήμαρχο της ΝΑΝΣ και τώρα ο λόγος στο Δήμαρχο του Μπουργκά, στον κύριο Νικόλ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού, Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω, διότι μου δίνετε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε και εμείς ε, σε ένα τέτοιο βήμα. Ε, για μένα με την ιδιότητά μου ως δήμαρχος αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία να έρθω σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ μέρους ε, των συμπολιτών μου. Η σημερινή μου συμμετοχή εδώ αποτελεί πραγματική δημοκρατία στην πράξη, αλληλεγγύη στην πράξη. Οι βασικές ευρωπαϊκές αξίες συνάδουν και με τη δική μου την ε, ιδέα να σας παρουσιάσω την κατάσταση ε, μιας πόλης ε, μεσαίου μεγέθους στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης η οποία προσπαθεί να ζήσει με υψηλούς στόχους βιώσιμα και προσπαθώντας να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών της. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μου και έχει συγκεκριμένες προκλήσεις. Και ως ε, Μητρόπολη πρέπει να κάνουμε περισσότερα προκειμένου να αναγνωριστούμε ως ε, μια ε, καλή πόλη για να ζει και να εργάζεται κανείς. Ε, προσπαθούμε να προσελκύσουμε άμεσες ξένες επενδύσεις και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να επενδύσουμε σε κοινωνικό κεφάλαιο. Βρισκόμαστε στις ακτές ε, του Ευξήνου Πόντου, στη νότια ακτή, ε, πολύ καλές κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Δυστυχώς όμως, τις τελευταίες δεκαετίες η πόλη αναπτύχθηκε περισσότερο ως κέντρο βαριάς βιομηχανίας και όχι πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο και προσπαθούμε τώρα να επανεξετάσουμε τους στόχους μας ώστε να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη, ε, ισορροπημένη αστική περιοχή και να μπορέσουμε να έχουμε ε, μια ανταγωνιστική ε, αστική κοινότητα. Και πλέον αρχίζουν να μας αναγνωρίζουν και περισσότερο στο χάρτη. Το 2014 είχαμε 36% αύξηση ε, τουριστικών επισκέψεων σε σχέση με το 2007. Γίνονται πολλά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία επίσης. Υπάρχει ε, μια πολύ καλή εταιρική σχέση με την ε, τοπική επιχειρηματική κοινότητα και η διοίκηση της πόλης προσπαθεί να παράσχει όλα τα απαραίτητα κίνητρα ε, θεωρούμε όλο ένα και περισσότερο ότι δεν είμαστε μια πόλη στην άκρη της Ευρώπης, αλλά μια πόλη στο κέντρο της Ευρώπης. Το γεγονός ότι υπάρχει καλή διασύνδεση και υποδομές ε, είναι ε, βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξή μας σε έναν διευρωπαϊκό διάδρομο. Το 2014 το αεροδρόμιό μας υποδόχθηκε πάνω από 2,5 εκατομμύρια τουρίστες και ε, η αύξηση εμπορευμάτων από θαλάσσεις ε, ε, ήταν πάρα πολύ καλή. Για το διάστημα 2007-2014 εγκρίθηκαν 37 προγράμματα για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από τα επιχειρησιακά μας προγράμματα. Από αυτά, τα 21 προγράμματα έχουν περατωθεί επιτυχώς. Άνω του 73% ε, των πληρωμών έχουν εκτελεστεί. Αλλά αυτά δεν είναι παρά ε, στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία. Η ποιότητα είναι πολύ πιο σημαντική από την ποσότητα και ο στόχος είναι να υπάρχουν συνέργειες στις επενδύσεις. Όπως βλέπετε υπάρχουν τα διάφορα στοιχεία ε, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του επενδυτικού περιβάλλοντος και ε, βασιζόμαστε και σε εθνική χρηματοδότηση για τα προγράμματά μας. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε στοιχεία τα οποία έχουμε ήδη επιτύχει ώστε να έχουμε πολλαπλά αποτελέσματα. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σημαίνει ευφυή, βιώσιμη ε, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς που σημαίνει ε, ότι ε, στην πράξη θα πρέπει να επενδύσουμε σε υποδομές, περιβάλλον, οικονομική ανάπτυξη, πολιτισμό είναι και ένα στοιχείο ε, για να νιώθουν καλύτερα και οι συμπολίτες μας. Βλέπετε εδώ στις φωτογραφίες κάποιες από τις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται, ε, κάποια από τα βασικά μέσα που διαθέτει η πόλη. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί με ε, καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. Και πάλι όπως σας είπα ε, το θέμα δεν αφορά την ποσότητα, αποτελεί ένα νέο ορίζοντα για την εκπλήρωση των φιλοδοξιών μας. Η πόλη μας είναι, ε, μάλλον κάθε πόλη είναι ε, όσο μεγάλη τις επιτρέπουν οι φιλοδοξίες της, αν μου επιτρέπετε να παραφράσω λίγο ε, μια γνωστή ρίση. Και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε επιτύχει έχουν αλλάξει το πρόσωπο της πόλης μας. Γι' αυτό ακριβώς και οι στόχοι που έχουμε διατυπώσει για τη νέα προγραμματική περίοδο ε, από το 2014 έως το 2020 είναι να συνεχίσουμε την επιτυχία και φυσικά είναι και ακόμα πιο φιλόδοξα προγράμματα ε, για ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον, καλύτερη ποιότητα ζωής ε, με κατάλληλη ενεργειακή απόδοση διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς επίσης. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να στάθηκα στο ύψος της υπόσχεσής μου, να σας δώσω μια εικόνα της πόλης μου που βρίσκεται στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, αρκετά μακριά βέβαια από το κέντρο της ε, Ευρώπης, ε, αλλά είναι πιο κοντά από ό,τι φαίνεται. Και η υποστήριξη για αστικές κοινότητες όπως η δική μας από πλευράς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, η αστική διάσταση στις ευρωπαϊκές πολιτικές ε, είναι κάτι το οποίο ε, μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό και εμείς θεωρώ ότι αποτελούμε ζωντανό παράδειγμα ε, της όλης αυτής της πολιτικής. Η προστιθέμενη αξία ενός θεματολογίου είναι πρωτίστως το γεγονός ότι θα μπορέσουμε να υπερκερέσουμε την τομεακή διαφοροποίηση. Είναι μια ολιστική, ολοκληρωμένη προσέγγιση και για εθνικούς αλλά και για διεθνείς σκοπούς. Από πλευράς ευρωπαϊκών πόλεων ένα τέτοιο θεματολόγιο θα μας βοηθήσει να αναγνωριστεί ο πραγματικός ρόλος των πόλεων ως κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης. Και από τις πόλεις, στο εθνικό επίπεδο, μπορούμε να αναμένουμε ακόμα πιο επιτυχή προγραμματισμό και προσέγγιση για την καλύτερη εθνική ανάπτυξη. Τέλος, κατ' εξίσου σημαντικό, το αστικό θεματολόγιο θα επιτρέψει στις αστικές κοινότητες να μπορούν να έρχονται σε επαφή και ε, άμεσα με, τις, ε, με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να αναγνωρίζονται ως πλήρης εταίροι στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης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 Συνεχίσουμε στις 3 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.